Äh, Κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η συνεδρίασή μας. Σας καλωσορίζω, ελπίζω να περάσετε ωραία το μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα οι ανακοινώσεις και σας παρακαλώ να εγκρίνετε αυτά τα οποία συμφώνησαν, προτείνουν οι συντονιστές. για το ζήτημα νομική προστασία των συμφερόντων της κοινότητας. Η κυρία Γκρέσλε θα ετοιμάσει ένα σχετικό έγγραφο. Ελπίζω να συμφωνείτε. Ωραία. Για το θέμα των διαρθρωτικών ταμείων και συγκεκριμένα το κοινωνικό ταμείο ναι, εκεί πέρα είναι αρμόδιο το ΕΛΚ, το οποίο θα ορίσει έναν εισηγητή. Θα το καθορίσουμε, θα το κάνουμε με την πορφή μιας επιστολής γιατί βεβαίω αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων για την μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Ταμείου και δεν γίνεται αλλιώ, οπότε θα ορίσει έναν εισηγητή το ΕΛΚ θα κανονιστεί αυτό με μια επιστολή του Προέδρου. Κατόπιν για το ανεκτό ποστό κινδύνου είχαμε χτες ε, μια συζήτηση και είχαμε πει ε, και πρέπει να γίνουν επαφές με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου, κάτι το οποίο θα κάνει ο Πρόεδρος. Εγκρίνεται λοιπόν και αυτό. Τον Φεβρουάριο θα συζητήσουμε για το λεγόμενο peer review και αυτό γίνεται δεκτό για τις ε, ε, ειδικέ εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου εδώ μέχρι το Μάρτιο του 2009 αναμένουμε μια έκθεση για το πρόγραμμα δημόσιας υγείας Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007. Ε, το ΕΛΚ είναι εδώ πέρα που έχει αναλάβει αυτό το θέμα και θα ορίσει έναν εισηγητή. Και για τις υπόλοιπες ε, ειδικέ εκθέσεις ε, καταλήξαμε στα εξής. Θα επεξεργαστούμε, θέλουμε να επεξεργαστούμε όσο δυνατόν περισσότερες σε αυτή την περίοδο, αλλά βεβαίως κάποιες θα παραμείνουν Δεν θέλουμε να έρθει κάτι το, το Μάρτιο για να το αναλάβουμε θα πάει στο επόμενο κοινοβούλιο οπότε οι υπόλοιπε εκθέσεις έχουν μοιραστεί απλά τις αναφέρω, τις αναφέρω στα αγγλικά γιατί στα αγγλικά ειδική έκθεση 8-2008 πολλαπλή συμμόρφωση και αποτελεσματική πολιτική Γιάννου Σοτσκόφσκι. η 9 η ειδική έκθεση 9 του 2008 αποτελεσματικότητα της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον τομέα δικαίου, ασφάλειας και ελευθερίας ε, Μολδαβία, Ουκρανία και Λευκορωσία, η κυρία Λιούπτσεβα. Επίσης, Προσεχώς προβλέπεται άλλη μια έκθεση υπαριθμών 10-2008 αναπτυξιακή βοήθεια στις υπηρεσίες υγείας στην υποσαχάρη Αφρική. Κυρία Στάς, εισηγήτρια και επίσης η έκθεση μέσα προενταξιακής βοήθειας ΙΣΠΑ 2000-2006 και εδώ πέρα θα... Εδώ πέρα προτείνεται ο αντιπρόεδρος κ. Λιμπεράτσι από τους σοσιαλιστές. Οπότε Τα εγκρίνεται ή μάλλον έχετε ενημερωθεί για αυτά. Ωραία. Και τελευταίο σημείο, ανανέωση της Εποπτικής Επιτροπής του Όλαφ. Γνωρίζετε πως υπήρχαν κάποιες αποφάσεις με βάση την έκθεση Γκρέσλε, εν μέρη ανανέωση δηλαδή της εποπτικής αυτής επιτροπής που θα πρέπει να λάβει χώρα, οπότε θα έχουμε μια επιστολή, είχαμε η επιστολή του κυρίου Κάλλας και μετά ο κύριος Πέτερινγκ εξήγησε τη θέση του Κοινοβουλίου ως πρόεδρος και χτες είχαμε νομίζω μία απάντηση από τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν τον κύριο Κάλλας και η πρόταση των συντονιστών είναι να προσπαθήσουμε να συστήσουμε μία ομάδα εργασίας που θα αποτελείται από το Προεδρείο της Επιτροπής μας και την μόνιμη εισηγήτρια για τον Όλαφ, την κυρία Γκρέσλε. Έχετε εδώ πέρα μια παρατήρηση, όχι, εγκρίνεται, οπότε εγκρίνονται όλα. Σας ευχαριστώ όλες οι συστάσεις των συντονιστών και περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Πριν περάσουμε όμως στην ημερήσια διάταξη, επειδή μεταδιδόμαστε και στο διαδίκτυο ζωντανά, γιατί υπήρχε μια συζήτηση για το αν είμαστε στο Web TV ή όχι. Μιλάμε για την διαφάνεια, είμαστε μια επιτροπή που μας απασχολεί διαφάνεια. Πράγματι τις δύο αυτές ημέρες μπορεί να μας δει κάποιος από οπουδήποτε στον κόσμο και δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον το πρόσωπό μου για να φανεί οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά εν πάση περιπτώσει χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι στην τελευταία σειρά βρίσκεται ένας πρώην συνάδελφος εδώ πέρα, ο Φρέντι Μπλακ, τον οποίον θα ήθελα να καλωσορίσω και προσωπικά. Καλώς ήρθατε, Φρέντι Μπλακ, στην παλιά σας ε, επιτροπή. Ήταν ο Φρέντι Μπλακ ε, επίμακρον αντιπρόεδρος αυτής της επιτροπής. Καλώς ήρθατε λοιπόν στα παλιά σλιμέρια. Οπότε περνάμε στο σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης απαλλαγή 2007, απαλλαγή της Κομισιόν. Δεν χρειάζεται να σας πω ποιος είναι ο εισηγητής. Είναι ο κύριος Σοντή. Καλώς ορίζουμε την κυρία Χίμπνερ. Και αργότερα θα έρθει και ο κύριος Ποτότσνικ εδώ πέρα. Καλώς ορίζουμε επίσης ε, και τα δύο μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την κυρία Καριολάινιν και τον κύριο Νόβακ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Τον λόγο έχει πρώτα απ' όλα το ελεγκτικό συνέδριο. Κυρία Καλγιολουλάιτ, Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού, κύριε Επίτροπε, θα σχολιάσω τα σπουδαιότερα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης του συνεδρίου για την πολιτική της συνοχής στην Ένωση. Η πολιτική συνοχή έγκυται από τα τέσσερα διαθετικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχή. Το 2007 η χρηματοδότηση της κοινότητας για την συνοχή ήταν 42 δις ευρώ ή 36,9% των συνολικών πληρωμών του προϋπολογισμού 2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έλεγχη για πληρωμές όσον αφορά τα διαθωτικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και την νομιμότητα και νομοτυπία των προσωρινών πληρωμών από τα ταμεία για το 2007. Κατά τον έλεγχο λοιπόν η εξέταση έγινε και από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως έχετε υπόψη οι έλεγχοι στα κράτη-μέλη στοχεύουν στο να αναγνωρίσουν και σε σχέση με τις ε, επιμέρους πληρωμές προς τους ε, αποδέκτες ε, να δουν τι γίνεται. Το ελεγκτικό συνέδριο ανέλησε 16 προγράμματα στα κράτη-μέλη και 11 από αυτά τα συστήματα θεωρήθηκαν εν μέρει αποτελεσματικά, τρία μη αποτελεσματικά και δύο πλήρως αποτελεσματικά οι αδυναμίες για τις διαφορές ε, για, όσον αφορά τους για τις ε, αρχές διαχείρισης ήταν μη επαρκής έλεγχη καθημερινή για την πραγματικότητα των δαπανών. Έλλειψη τεκμηρίων και αδυναμίες όσον αφορά την διαδικασία προμηθειών ή αγορών σφάλματα τα οποία έγιναν όσον αφορά τις ε, καθημερινές, τους καθημερινούς ελέγχους. Αποτυχία να υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι για την λειτουργία των συστημάτων αυτών. Και το έργο των ε, ε, όσων εμπλέκονται θεωρείται αποτελεσματικό στις ε, περιπτώσεις που ανέφερα. Επίσης ε, το δεύτερο μέρος ελέγχου όσον αφορά τα προγράμματα συνοχής ε, στοχεύουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο του να μην υπάρχουν αποτελεσματικοί έλεγχοι στα κράτη-μέλη. Για να το πω πιο απλά, <clears throat> όχι τόσο πολύ τα επιμέρους φάρματα αλλά εκείνο το, τα συστήματα στα οποία οφείλεται η διολίστηση αυτή. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί αυτό όσον αφορά το πάγωμα των πληρωμών και τις ε, εφάπαξ ε, πληρωμές κατά αποκοπή που οφείλονται στα κράτη-μέλη αλλά όχι σε επιμέρους προγράμματα. Η Επιτροπή εν μέρη εντοπίζει μη αποτελεσματικού ελέγχου στα κράτη-μέλη μέσω των ελεγκτικών δραστηριοτήτων τη. Ανέλησε 22 τέτοιου ελέγχου τη Επιτροπής ε, το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά το πεδίο τη συνοχή. Στην πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων οι έλεγχοι είχαν σχεδιαστεί και έγιναν αποτελεσμα... επαρκώ. Έτσι λοιπόν για το 2007 για ε, την ετήσια έκθεση της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζεται ένα μέγεθος πολύ ανώτερο από εκείνο του 2006, πράγμα που καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τις αναλύσεις του ίδιου του ελεγκτικού συνεδρίου. Υπάρχουν και άλλες πτυχές στην εποπτική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι τακτικές δαπάνες θα καλύπτουν, θα ανακτώνται από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό πρέπει να συλλέξει, να αναλύσει και να εποπτεύσει αυτή τη διαδικασία Επιτροπή. Όμως, εν η Επιτροπή για το 2007 ακόμα δεν ήταν σε θέση να αποδείξει ότι τα μεγέθη τα οποία παρουσιάζουν λαμβάνουν υπόψη όλες τις συναλλαγές των κρατών μελών και για την ε, ε, δημοσίευση και σύγκριση με τις δημόσιες δαπάνες. Έτσι λοιπόν για το 2008 θα πρέπει σίγουρα να επιτευχθούν βελτιώσεις. Ωστόσο ο αποτελεσματικός έλεγχος δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αποτελεσματική έλεγχη είναι μέσα, εργαλεία για να αποφύγουμε σφάλματα Στρέφομαι τώρα στην εξέταση από το ελεκτικό συνέδριο των συναλλαγών. Εξέτασε 180 τέτοιου είδους ε, προσωρινές συναλλαγές που έγιναν το 2007 για την περίοδο 2000, από την περίοδο 2000-2007 46% των σχεδίων ή προγραμμάτων ήταν χωρίς φάλματα ε, σωστά ε, εξοφλήθηκαν και, και δεν είχαν ε, επίσης και σφάλματα συμμόρφωσης. Όσον αφορά το 2006 το ποσοστό αυτό ήταν 31% για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Εδώ υπήρξαν σημαντικά σφάλματα για το, η έλλειψη στοιχείων όσον αφορά και επίσης και τις δαπάνες προσωπικού και μη επιλέξιμα κόστη είχαν ε, ε, τη ρίζα τους σε σφάλματα. Έτσι και όπως για πέρσι υπολόγισε το ελεγκτικό συνέδριο το ποσοστό ε, υπερβολικών δαπανών. Είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν θα έπρεπε να είχε επιστραφεί ή ανακτηθεί. Και για φέτος εκτιμά το Συμβούλιο ότι το συνολικό όριο για την ε, περίπτωση αυτή είναι 11%. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνουν ότι το ελεγκτικό συνέδριο κατά 95% πιστεύει ότι σφάλματα σε σχέση με τέτοιου είδους συναλλαγές θα είναι ή 11% ή παραπάνω. Επίσης και σοβαρότερα σφάλματα δεν έχουν ε, ποσοστοποιηθεί ακόμα, αποκλείονται από αυτούς τους λογαριασμούς. Έτσι λοιπόν 11% είναι το ποσοστοποιήσιμο ε, σφάλμα όσον αφορά τους ακριβείς λογαριασμούς. Τώρα, η, ε, ως ήθιστε υπενθύμησε, δεν υπάρχει απλή απάντηση στο θέμα αν αυτά τα χρήματα χάθηκαν. Το μόνο το οποίο είναι σαφές είναι ότι ενώ δαπανώνται, τα σφάλματα έναντι νομοτυπίας και νομιμότητας ε, ήταν δεδομένα και πράγματι είναι απίθανο τα κονδύλια αυτά να μπορέσουν να ανακτηθούν από τους τελικούς ε, εποφελούμενους αποδέκτες. Είναι περισσότερο πιθανό να αντικαταστήσουν τα κράτη-μέλη τα μη ορθώς καταβεβλημένα ποσά και να αντισταθμίσουν με νέα από τα νέα ποσά. Μια και βρισκόμαστε στην φάση που κλείνει η περίοδος 2000-2006 ε, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτή η φάση έχει κέρια σημασία για την τελική έκβαση των δαπανών των ταμείων αυτών. Τέλος, δύο σύντομα, ένα σύντομο σχόλιο για τις συστάσεις του ελληνικού συνεδρίου. Όπως πάντα, όταν είναι άκρημα τα σφάλματα, υπάρχει αυτόματη σύσταση να διασφαλιστεί ότι η διαχείριση και η ε, σωστή εφαρμογή θα διασφαλίζεται όπως πρέπει γνωρίζει το Συμβούλιο και το έχει αναφέρει αυτό και στην ετήσια έκθεση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος για ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης για τα κράτη-μέλη και για τους τελικούς αποδέκτες. Γι' αυτό λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, το Συμβούλιο συνέστησε και Τώρα, αναφέρομαι από την απάντηση προς την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ε, μεταρρύθμιση τη δημοσιονομική συνέστησε το λεκτικό συνέδριο οι πολιτικές αρχές να είναι έτοιμες, θα πρέπει να είναι έτοιμες μέσα στο πλαίσιο μιας θεμελιώδους μεταρρύθμισης του προϋπολογισμού δημοσιονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβληματιστούν τι θα γίνει με την πολιτική δαπανών στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστούμε και για αυτές τις ε, ακριβείς ε, συνοψίσεις, ε, περιλήψεις μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είναι θέματα τα οποία έχουν σημασία για μας σας και πρέπει να μιμηθούμε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την κυρία Καλιουλάκη για την ισορροπημένη παρουσίαση της, του σχετικού κεφαλαίου της ε, ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και βεβαίως το ότι αυτό ακόμα δεν αντικατοπτρίζεται σε μια σοβαρή μείωση του ποσοστού σφαλμάτων. Η Κομισιόν έχει δείξει πω παίρνει πολύ σοβαρά τι ευθύνε τη όσον αφορά τη διαχείριση του υπερπολογισμού. Πέρυσι τον Φεβρουάριο υιοθετήσαμε το σχετικό σχέδιο δράση για τι δράσει αυτέ λόγω των πολύ σαφών μηνυμάτων που λάβαμε από την Επιτροπή σα στην απαλλαγή του 2006. Πώς θέλατε δηλαδή άμεση δράση για να έχουμε μικρότερο ποσοστό σφαλμάτων σε αυτό τον τομέα πολιτικής. Νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε. Η τελική έκθεση της Κομισιόν θα υιοθετηθεί στις 3 Φεβρουαρίου και δείχνει πως οι περισσότερες από τις 37 αυτές δράσεις έχουν ολοκληρωθεί και η Κομισιόν ε, διαχειρίζεται πάρα πολύ σφρίγγυλα αυτή την πολιτική. Να σας αναφέρω το ότι το 2008 υιοθετήσαμε 10 αποφάσεις για αναστολή πληρωμών γιατί τα κράτη-μέλη δεν είχαν επαρκή συστήματα ελέγχου. Το 2007 είχαμε μια τέτοια απόφαση. Για τις δημοσιονομικές διορθώσεις υιοθετήσαμε 26 τέτοιε αποφάσει σε, σχέση, σε σύγκριση με, 26, με 16 το 2007 και το ποσό ανήλθε σε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2000-2006 για ΕΤΠΑ και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και μαζί με την ε, προηγούμενη περίοδο φτάνει στο 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή έχουμε ένα πενταπλασιασμό σε σύγκριση με το 2007 και αυτό το οποίο προγραμματίζουμε είναι λίγο πολύ 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης παρακολουθούμε συστηματικά όλα τα λάθη τα οποία βρίσκονται είτε από τον όλα αυτή στις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά η αφετηρία του... άνω του 80% των διορθώσεων είναι η έλεγχη της ίδιας Κομισιόν. Εκτιμώ πως σήμερα κυρίως μας, ε, και αντιλαμβάνομαι πως σήμερα μας απασχολεί κυρίως το 2007 και υπάρχουν κάποια θετικά νέα στην έκθεση του Ενεκτικού Συνεδρίου. Υπάρχει μια καλύτερη γενική αξιολόγηση της λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου και εποπτείας. Για πρώτη φορά έχουν πάρει βαθμολογία κίτρινη, δηλαδή εν μέρει αποτελεσματικά τα συστήματα ελέγχου και της Κομισιόν και των κρατών μελών. Υπάρχει σαφή βελτίωση λοιπόν των συστήματων διαχείρισης και ελέγχου και όπως είπε και η κυρία Καλιλέιτ, από τα 16 προγράμματα που έλεγξε το ελεγκτικό συνέδριο, μόνο σε τρία το σύστημα θεωρήθηκε ανεπαρκές. Στην περίπτωση του 6 είχαμε 13 από τα 19 συστήματα που κορυφθήκαν αναποτελεσματικά καλύτερα είναι τα πράγματα στο ποσοστό των έργων που θεωρήθηκαν ότι δεν υπάρχουν, δεν έχουν λάθη. Κάτι το οποίο αυξήθηκε κατά 15% σχέση με το 2007. Επίσης, ψηλότερη βαθμολογία δίνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριότητας ανα γενική διεύθυνση. Κάτι το οποίο σημαίνει πως δεν υπάρχουν πλέον ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στην Κομισιόν και το ελεγκτικό συνέδριο στην αξιολόγησή του. Οπότε η τάση πάει προ σωστή κατεύθυνση, κάτι το οποίο δείχνει πω οι τη Κομισιόν τα τελευταία χρόνια μέσω όλων των σχεδίων δράσεων, ε, εκπαίδευση, ε, όλα αυτά αποφέρουν αποτελέσματα. Αλλά να τονίσω ξανά πω το ποσοστό σφάλματο 11% είναι σαφώ πολύ ψηλό. Οπότε πώ θα διασφαλίσει η Κομισιόν πώ οι βελτιώσει αυτέ του συστήματο θα μεταφραστούν σε ένα σαφώ χαμηλότερο ποσοστό σφάλματο. Υπάρχουν πέντε δράσει που Έχουμε ξεκινήσει. Πρώτα απ' όλα έχουμε τη σκληρή προσέγγιση για την αναστολή και τις ε, δημοσιονομικέ διορθώσεις που είναι κίνητρο για τα κράτη-μέλη να έχουν αποτελεσματικούς πρωτοβάθμιους ελέγχους. Δεύτερον, Έχουμε αυστηρούς ε, ελέγχους για το 2007-2013. Τρίτον, θα έχουμε μια αυστηρή διαδικασία κλεισίματος για τα προγράμματα 2000-2006. Τέταρτον, θα φροντίσουμε τα κράτη-μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές αναφέρονται στις αιτήσει εκθέσεις. Και έχουμε νέες κατευθύνες γραμμές για το 2008 επίσης θα επανέλθουμε τον Μάρτιο για να σας πούμε τα αποτελέσματα των ετήσιων εκθέσεων του 2008. Να σας διαβεβαιώσω πως η Κομισιόν συνεργάζεται ενεργά με τα κράτη-μέλη που εθελοντικά είχαν συμφωνήσει να κάνουν εθνικές δηλώσεις γιατί θεωρούν πως αυτή η δέσμευση από πλευράς κρατών μελών μπορεί να βοηθήσει την καλύτερη διαχείριση επιτόπου. Πέμπτον, έχουμε αναλάβει δραστικά μέτρα προς την πλευρά της απλοποίησης. Υπάρχει μια γενική συμφωνία πως η υποϋποκότητα των κανόνων ε, προκαλεί το υψηλό ποσοστό σφαλμάτων. Επίσης, έχω συστήσει εγώ μια ομάδα ειδικών για να δει τι μπορεί άλλο να γίνει βραχυπρόθεσμα, αλλά είναι σαφές πως η Κομισιόν δεν θα υιοθήσει κάποιες αλλαγές για να γίνουν ασθενέστεροι έλεγχοι στην περίοδο 2007-2013. Τέλος, το ποσοστό του ανεκτού σφάλματος, κάτι που είναι σημαντικό για τα διαρθρωτικά μέτρα για δύο λόγους. Γιατί είναι μια πολιτική που έχει πολύ μεγάλο εγγενή κίνδυνο λόγω του επενδυτικού της χαρακτήρα, γιατί μιλάμε για επένδυση σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και οι δράσει αναπτύσσονται σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Κατόπιν πρόκειται για πολυετή πολιτική που αναπτύσσεται σε βάθος χρόνου. Οπότε το ετήσιο ποσοστό σφαλμάτων είναι μάλλον υψηλότερο από ό,τι στο τέλος του προγράμματος. Επίσης παρακολουθούμε συστηματικά, καταλήγοντας κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, η πολιτική συνοχή είναι μια πολιτική κλειδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τονίστηκε και από το σημαντικό ρόλο που παίζει το πακέτο ανάκαμψης. Γι' αυτό οι προσπάθειέ μα να ενισχυθεί ο έλεγχο και να έχουμε μείωση του ποστού σφάλματος είναι τόσο σημαντικέ. και η έκθεση του Δικαστηρίου για το 2007 περιέχει ενθαρρυντικά σημεία προόδου και με τη βοήθεια και της Επιτροπής σας Κομισιόν έλαβε σοβαρά μέτρα για την εφαρμογή της σχεδίου δράσης που έχουν στο αποτέλεσμα θετικά αποτελέσματα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Äh, Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω τον λόγο στον συγκεκριτή να πω πως χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων κ. Σούλμπριχτ είναι εδώ και η συντονίστρια των Σοσιαλιστών κυρία Κρέλ στην Επιτροπή αυτή, οπότε νομίζω πως θα αποκτήσει και περισσότερη ουσία η συζήτησή μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Τον λόγο έχει ο γενικός μας συγητής, ο κ. Σοντή, για την λεγόμενη διαδικασία ping-pong. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα πρώτα μου λόγια θα απευθυνθούν στην Επίτροπο για να ευχαριστήσω για τη συνεισφορά της στην συνεδρία εργασίας. Θέλω να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο για την έκθεσή της που μου επιτρέπει, μας επιτρέπει να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Κοιτάστε, για λόγους ε, πένθους ε, σε ένας φίλος μου θα χρειαστεί να επανέλθω στην... θα πρέπει να, να γυρίσω στην πατρίδα μου και θα με αντικαταστήσει συνάδελφος. Κυρία Επίτροπε, πόσες πληρωμές κάνετε εσείς ε, στις πολιτικές των οποίων έχετε την αρμοδιότητα, έχετε την πολιτική συνοχή, έχετε τη γεωργία και άλλες πολιτικές, έχετε όμως τις μεγάλες πολιτικές, πόσες πληρωμές κάνετε το χρόνο όχι, όχι το ποσό, όχι το συνολικό ποσό, αλλά πόσες πράξεις πληρωμής. Να σας απαντήσω τώρα. Ναι. Γενικά μπορώ να πω πως η Κομισιόν κατά μέσο όρο κάνει τρεις ενδιάμεσες πληρωμές ανά πρόγραμμα κάθε έτος, δηλαδή γύρω στις 1600 πληρωμές και αντιπροσωπεύουν τις ε, πλήρωμες σε όλα τα ανοιχτά έργα. Δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό, είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή. Για το ΕΤΠΑ κρίνουμε πως ε, συνολικός αριθμός είναι 700.000 ε, και για το ΕΚΤ αν λάβετε υπόψη το μέγεθος των έργων που είναι σαφώς μικρότερο είναι οπωσδήποτε λιγότερε πληρωμέ, αλλά ίσω οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση ξέρουν τον ακριβή αριθμό. Εφτακόσες χιλιάδες πληρωμές, πράξεις πληρωμής το χρόνο, κατάλαβα καλά. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Διευθυντή να απαντήσει. Ευχαριστώ η Κομισιόν ε, καταβάλει ενδιάμεσε πληρωμές στα κράτη-μέλη αναπρόγραμμα. πρόγραμμα. Όπως είπε η κυρία Επιτροπός, κατά μέσο όρο ε, λαμβάνουμε τρει αιτήσει για ενδιάμεσε πληρωμές αναπρόγραμμα, πρόγραμμα, ανά έτος. Και καθώς υπάρχουν 545 προγράμματα για όλα τα διαρθρωτικά ταμεία, αυτό σημαίνει πως ε, αναέτος η Κομισιόν ε, κάνει γύρω στις 1.600 ενδιάμεσες πληρωμές προς τα κράτη-μέλη στα προγράμματα. Αλλά πίσω από αυτό κρύβονται τα μεμονωμένα έργα του κάθε προγράμματος. Οπότε οι πληρωμές προς τα κράτη-μέλη αφορούν ουσιαστικά καταβολές στα συγκεκριμένα έργα και σε επίπεδο Κομισιόν δεν έχουμε λεπτομέρειες όλων των έργων γιατί αυτό είναι κάτι που γίνεται σε επίπεδο κράτους μέλους εντός του προγράμματος. Αλλά Αποστολή υπολογίζουμε για το ΕΤΠΑ πως υπάρχουν γύρω στις 700.000 έργα που είναι ανοιχτά μάλλον ανοιχτά να πάει στιγμή είναι τα μισά από αυτά και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι πάνω από ένα εκατομμύριο οπότε πίσω από αυτές οι ενδιάμεσες πληρωμές όπως σας είπα υπάρχουν αυτές οι, οι πληρωμές που γίνονται σε πάνω από ένα εκατομμύριο έργο, πιθανότατα. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Εσείς ε, κάνετε πληρωμές, ε, καταβάλλετε δηλαδή τις πληρωμές στα κράτη-μέλη και μετά τα κράτη-μέλη ε, με καταμερισμένη διαχείριση κάνουν και με τη σειρά τους και αυτά τις πληρωμές. Τώρα, βάσει των ελέγχων, δηλαδή έγιναν 180 έλεγχοι για να, ελεγχ, για να ε, ελεγχθούν 700.000 πληρωμές. Το θεωρείτε επαρκές? Ναι. αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι τεχνικό, σύμφωνα με το πρόγραμμα διασφάλισης ε, του ελεγκτικού συνεδρίου χρειαζόμαστε γύρω στις, ε, ένα μέγεθος δείγματος γύρω στο 180 για να έχουμε μια διασφάλιση ότι έχουμε μηδενικό σφάλμα. Οπότε ναι, μπορούμε να φτάσουμε σε μια λογική, σε μια θετική ε, γνωμοδότηση. Έτσι λειτουργεί το μοντέλο διασφάλισης για το πώς καθορίζουμε το μέγεθος του δείγματος. Οπότε αν είμαστε πεπισμένοι από την παρελθούσα εμπειρία πως το αποτέλεσμα μάλλον θα είναι αρνητικό, μπορούμε να κρίνουμε με πολύ μικρότερο ύψος δείγματος, να αποδείξουμε στατιστικά πως υπάρχουν ε, μικρότερα, λιγότερα λάθη. με το 180 είμαστε 95% σίγουροι πως το χαμηλότερο ποσοστό σφάλματος είναι 11% για το 2007. Αυτό επαληθεύεται και από τη μεθοδολογία που ακολουθείται διεθνώς. Merci, euh, merci, madame. Ευχαριστώ κυρία μου. Εγώ θέλω να επανέλθω στη διαδικασία, δηλαδή στην τριετή έκθεση για το σχέδιο δράσης που μας παρουσιάσατε κυρία Επίτροπε σχετικά με το ποσοστό λάθος 12% για το 2006 έχει κατέβει στο 11% φέτος. Εσείς ε, τι, τι, τι, τι εντύπωση έχετε για τα αποτελέσματα, για τις επιπτώσεις του σχεδίου δράσης ε, πώς ερμηνεύετε τη μείωση του ποσοστού και ποια είναι η προσωπική σας άποψη για την εκτίμηση του ελεκτικού συνεδρίου που εκτιμά ότι το 11% των καταβεβλημένων ποσών δεν θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί. Λοιπόν, εσείς πώς το βλέπετε αυτό, έγιναν 180 έλεγχοι για 700.000 πληρωμές. Η Κομισιόν όπως και όλοι, θεωρεί απαράδεκτο το ποσοστό σφάλματος 11%. Γι' αυτό έχουμε στόχο να το μειώσουμε. Γι' αυτό υιοθετήσαμε το σχέδιο δράσης με πολύ συγκεκριμένο στόχο. Να επικεντρωθούμε σε μια σειρά δράσεων που τελικά θα μειώσουν το ποσοστό. Και όπως κατέστησα σαφές στην αρχική μας ομιλία, το έχουμε επιτύχει αυτό αυτό το οποίο είχαμε θέσει δηλαδή ως στόχο και θεωρούμε ότι έχουμε πρόοδο στον στρατηγικό στόχο της μείωσης του ποσοστού σφάλματος. Επίσης θα έλεγα πως σήμερα σε αυτή τη φάση γνωρίζουμε τους βασικούς τύπους σφάλματος και άρα μπορούμε να επικεντρωθούμε εκεί. Παραδείγματο χάρη στις διαδικασίες δημοσίων προμηθειών που είναι το βασικό είδος σφάλματος στην πολιτική και επιτόπου στα κράτη-μέλη έχουμε κανονίσει μια σειρά σεμιναρίων για να υπάρχει ενημέρωση για τις απαιτήσει και για να κινητοποιηθούν τα κράτη-μέλη να κάνουν περισσότερα όσον αφορά την κατάρτιση και την ενημέρωση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο επίσης. Συνιστούμε στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ανάλογο επίπεδο διορθώσεων για τις παρατυπίες με αυτό της Κομισιόν. Επίσης, συμφωνούμε με το συνέδριο πως η βασική πηγή ε, σφαλμάτων είναι η καθημερινή διαχειριστική έλεγχη γι' αυτό και έχουμε επικεντρωθεί εκεί και είχαμε μια σειρά στοχευμένων ελέγχων των φορέων διαχείρισης και σεμινάρια όχι μόνο για, τους, για τις αρχές διαχείρισης που παραδοσιακά είχαμε, αλλά και για τους φορείς πιστοποίησης. Ένα σεμινάριο με τον κύριο Μπες ε, που ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και σημαίνουμε επίσης πως ε, τα σφάλματα αφορούν παραβιάσεις κάποιων όρων της χρηματοδότησης και κάποιες είναι πιο σοβαρές αλλά δεν τίχτε ζήτημα του να μην ξέρουμε που πήγαν τα λεφτά μόνο δύο από τα 180 έργα που έλεγξε το συνέδριο είχαν υποψία απάτης και γνωρίζετε πως τα νούμερα του Όλαφ ε, υπολογίζουν το επίπεδο απάτηση στο 0,1% των ε, δαπανών και μιλάμε πάλι για υποψία δαπανής οπότε αν πάμε στις πραγματικές περιπτώσεις ε, θα είναι ακόμη χαμηλότερο Μπορώ να σας πω για το σχέδιο δράσης. Αναλάβουμε λοιπόν όλες αυτές τις δράσεις που επικεντρώνονται κυρίως σε αυτές τις περιοχές, σε αυτούς τομείς ανισχύες και κινητοποιήσαμε νομίζω και τα κράτη-μέλη να εμβαθύνουν αυτές τις δραστηριότητες. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε σε καλό δρόμο και αυτό με κάνει να έχω εμπιστοσύνη πως θα συνεχίσουμε να συνεισφέρουμε στο να συνεχίσει να πέφτει το ποσοστό σφάλματος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εγώ δηλαδή θα συγκρατήσω από την όλη σας απάντηση ότι θεωρείται απαράδεκτο το 11%, το θεωρείται πολύ ψηλό, αλλά συμφωνείτε σε αυτήν τη διαπίστωση. Δηλαδή, ότι το 11% του συνολικού ποσού που καταβλήθηκε δεν έπρεπε να, γίνει, να, να καταβληθεί. Και λέτε ότι θα έπρεπε να μειωθεί αυτό το ποσοστό. Αναγνωρίζετε βέβαια ότι δεν υπάρχει απάτη. Ο εισηγητής για την απαλλαγή, ο κύριος Γιώργενσεν, πέρυσι, ζητούσε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε, να γίνεται μία γενικότερη ποιοτική αξιολόγηση για τη γεωργία, την αλία και τις πολιτικές συνοχής. Δεν έχει γίνει αυτή η αξιολόγηση. Θα την φέρετε εδώ στο κοινοβούλιο τελικά, θα την υποβάλλετε. Θεωρείτε ότι αυτές οι αιτήσιες εκθέσεις που γίνονται κάθε χρόνο βελτιώνουν την κατάσταση στον έλεγχο του προπολογισμού. Εργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη κατά τα τελευταία δύο χρόνια μπορώ να πω για να διασφαλίσουμε ότι οι ετήσιες περιλήψεις θα παρέχονται και για πρώτη φορά δόθηκαν πέρυσι αλλά για εφέτος εκδώσαμε νέες κατευθυντήρες γραμμές σε σημειώσεις ε, το Δεκέμβριο πέρσι για να βελτιωθεί η ποιότητα και η χρησιμότητα των εθνικών αυτών συνόψεων ή περιλήψεων για να είναι συμβατές ε, συγκρίσιμες και να είναι χρήσιμες για τα κράτη-μέλη και σε εμά, για εμά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για την Ευρωβουλή και το Ελεγκτικό Συνέδριο ως πηγή πληροφοριών. Μπορεί να θυμόσαστε ότι δεν ήταν εύκολο το εγχείρημα αυτό επειδή το 2007 ενώ πιστεύαμε ότι θα δεσμευόντουσαν τα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν, υπήρχε μια πολύ αρνητική αρχική αντίδραση από τα κράτη-μέλη σε σχέση με την απόφαση του Συμβουλίου. Ε, είπαν τα κράτη-μέλη ότι η απόφαση του Συμβουλίου για την απόφαση αυτή για το δημοσιονομικό κανονισμό δεν καλύπτει την περίοδο 2000-2006. Δεν υποχρεώνει, με συγχωρείτε, τα κράτη-μέλη να παράσχουν τις ετήσιες περιλήψεις ή συνόψεις, αλλά μετά από πολλή δουλειά που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σιγά σιγά τα κράτη-μέλη συμμορφώθηκαν και όλα εκτός ενός είχαν στείλει τέτοιου είδους περιλήψεις που κάλυπταν τις ελάχιστες αναγκαίες προϋποθέσεις. Αυτό είναι το θέμα το σημαντικό για μας, διότι θεωρούμε ότι μπορούν να υποβάλλονται από τα κράτη-μέλη πολύ σε μεγαλύτερο βάθος ε, περιλήψεις ε, συνοπτικά, με πολύ μεγαλύτερο βάθος ανάλυσης υπό τους όρους των συντελεστών των παραγόντων που βρίσκονται πίσω από τους ελέγχους. Όχι απλά και μόνο μια παρήθμιση των ελέγχων που έγιναν κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Γι' αυτό σε αυτές τις νέες κατευθυντήρες γραμμές στο σημείωμα στην ανακοίνωση ζητούμε από τα κράτη-μέλη να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ανάλυση αυτή στις ε, περιλήψεις τους και για την, ε, το πιστοποιητικό την δήλωση αξιοπιστίας ε, Statement of Assurance. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από τα κράτη-μέλη από τις αιτήσει περιλήψεις να κάνουν κάτι παραπάνω από μία, ας το πω έτσι, ένα συνονθήλευμα, μία παρήθμιση κάποιων πληροφοριακών στοιχείων. Και από πλευράς του Διευθυντού μας απευθύνθηκε επιπρόσθετα σημείωση προς τα κράτη-μέλη ενισχύοντας περισσότερο αυτό το μήνυμα και ελπίζουμε ότι εφέτος θα πάρουμε όχι μόνο την περίληψη αυτών των πληροφοριακών στοιχείων, αλλά θα έχουμε και μια ανάλυση πώς δηλαδή λειτουργούν αυτά τα συστήματα στο επίπεδο των κρατών μελών και θα έχουμε και μια διάγνωση των προβλημάτων που διαπιστώνονται και τις λύσεις που θα μπορούν να ακολουθηθούν σε σχέση και με τις ευέλτιστες πρακτικές ε, όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Επίσης η δήλωση του βαθμού αξιοπιστίας ε, όσον αφορά τα όσα μπορούν να απορρεύσουν από αυτό το σύστημα για τα κράτη-μέλη. Ευελπιστούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτό και εργαζόμαστε για να βελτιωθεί η ποιότητα και η χρησιμότητα και για μας και για τους άλλους που εμπλέκονται για αυτές τις περιλήψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Πιο συγκεκριμένα και για την κριτική που γίνεται στα κατάσταση στα, σε ορισμένα κράτη-μέλη, στην έκθεση του 2007 που μοιάζει πολύ με εκείνη του 2006, ο Γενικός Διευθυντής της Περιφερειακής Πολιτικής σχετικά με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θέτει μία επιφύλαξη για 10 κράτη-μέλη και για 51 προγράμματα Interreg. Και για το Ταμείο Συνοχής θέτει επιφυλάξεις για 5 κράτη-μέλη. Πολλά μέτρα ελήφθησαν το 2007 2008 για να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς αυτό το θέμα της καταμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη-μέλη. Μπορείτε σύντομα να μας αναφέρετε αυτά τα μέτρα και για τα κράτη-μέλη για τα οποία εξέφρασε ανησυχίες το ελεγκτικό συνέδριο, τι λέτε. Γιατί ανησυχούμε ιδιαίτερα για την μέτρια ποιότητα της καταμερισμένης διαχείρισης και τα μέτρια αποτελέσματά της. Οπότε αμφισβητούμε ήδη το, ε, το ίδιο το σύστημα της καταμερισμένης διαχείρισης. Θα ήθελα να ζητήσω από τον ε, κύριο Διευθυντή να ξεκινήσει την απάντηση. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, το βασικό μέσο που έχουμε αυτή τη στιγμή στην διάθεσή μας στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης είναι αυτό το οποίο θα έλεγα μια στρατηγική push and pull. Από τη μία πλευρά αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο χρόνια είναι να ενημερώσουμε τα κράτη-μέλη το τι απαιτεί η νομοθεσία και να εξηγήσουμε για το πώς μπορούν να εκπληρώσουν αυτές τις απαιτήσει από την άλλη πλευρά. Έχουμε αλλάξει την προσέγγιση μας μετά την περσινή συζήτηση και έχουμε αλλάξει προσέγγιση όσον αφορά την αναστολή και διόρθωση των πληρωμών. Και τώρα η δράση μας είναι πολύ πιο γρήγορη από ό,τι στο παρελθόν. Κάτι το οποίο ήδη φαίνεται στα νούμερα του 2008. Όσον αφορά τώρα τους δικούς μας ελέγχους προσπαθούμε να στοχεύσουμε το ελεγκτικό μας έργο σε εκείνες τις διαχειριστικές αρχές όπου βλέπουμε τον υψηλότερο κίνδυνο με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από διάφορες πλευρές είτε από παλιότερους δικούς μας ελέγχους εν μέρη από το ελεγκτικό συνέδριο εν μέρη από άλλες πηγές προσπαθούμε να στοχεύσουμε το έργο μας εκεί όπου θεωρούμε ότι είναι ψηλότερος ο κίνδυνος. Με τη στρατηγική αυτή που έχει ενισχυθεί το, κατά το 2008, οφείλω να πω στο επίπεδο του, του ποσοστού σφάλματος δεν είναι σαφή ακόμα τα αποτελέσματα και προσωπικά οι προσδοκίες μου είναι όσον αφορά την περίοδο 2000-2006 θα δούμε διαφορετικά θα έχουμε αποτύχει, μία βελτίωση στο επίπεδο κλεισίματος των προγραμμάτων που ξεκινάει αυτή τη στιγμή και πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε τις δικές μας εκτιμήσεις στο Κοινοβούλιο για τον κίνδυνο που παραμένει μετά το κλείσιμο για να δούμε κατά τη διάρκεια της πολιτούς αυτής της διαδικασίας το τι έχει γίνει. Και τις προσδοκίες μας μετά το κλείσιμο ο κίνδυνος που απομένει πρέπει να είναι σαφώς χαμηλότερος από το ποσοστό σφάλματος που διαπιστώνουμε σήμερα όσον αφορά την περίοδο 2007-2013. Οπωσδήποτε ελπίζουμε να δούμε σαφώς ε, πιο σφιχτή έτσι προσέγγιση όπως υπάρχει στον κανονισμό και ελπίζουμε επέκταση σταδιακά στους ετσίους ελέγχους ε, το 2007-2013 όπου θα γίνει ο κύριος όγκος των πληρωμών αναμένουμε να πέσει το ποσοστό σφαλμάτων. Και τα δύο αυτά πράγματα θα είναι για εμάς τα βασικά κριτήρια με τα οποία θα μετρήσουμε την επιτυχία ε, της δουλειά μας. Εάν μου επιτρέπετε να προσθέσω δύο πράγματα για τις δράσεις μας για τη βελτίωση της κατάστασης ε, στα κράτη-μέλη μία δράση της Κομισιόν είναι οπωσδήποτε η προσπάθεια να αυξηθεί ο αριθμός των κρατών μελών με τα οποία έχουμε υπογράψει αυτές τις συμβάσεις ε, εμπιστοσύνη. Σε αυτή τη στιγμή έχουμε Αυστρία, Δανία, Εστονία, Πορτογαλία και ελπίζουμε και την Κύπρο να ε, υπογράψουμε επίσης άλλες δύο συμβάσεις με Δανία και την Ηνωμένο Βασίλειο Κάτι το οποίο οδηγεί κατά την άποψή μας προς μια γενικότερη βελτίωση του συντονισμού του ελεγκτικού έργου και δημιουργεί κάτι το οποίο είναι σημαντικό μια διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης και για τα κράτη εκείνα τα οποία δεν θέλουν να υπογράψουν μια τέτοια σύμβαση. Είναι μια σύμβαση που ισχύει όπως ξέρετε για την προγραμματική περίοδο 2000-2006 και θα διευκολύνει και το κλείσιμο, αλλά για την νέα περίοδο 2007-2013 τα βασικά στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας έχουν ενσωματωθεί στον κανονισμό. Οπότε θα συνεχίσει αυτό να έχει αποτέλεσμα. Και το δεύτερο μεταξύ όλων αυτών των πρωτοβουλειών που αφορούν εκπαίδευση και κατευθυντήριες γραμμές και τα λοιπά νομίζω για το 2007-2013 έχουμε ξεκινήσει αρκετά νωρίς νωρίτερα πριν ξεκινήσει όλη η περίοδος και δώσαμε κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη ακριβώς για τους πρωτοβάθμιους ελέγχους για τις αρχές πιστοποίησης για την αξιολόγηση συμμόρφωσης, για τις στρατηγικές ελέγχους, για το δείγμα, τη δειγματοληψία, επίσης για το μερικό κλείσιμο του 2007-2013, για, το... την περίπτωση στην οποία ξεπερνούσαμε τα ποσά στην περίπτωση των κοινωνικών ταμείων και όπως είπα για την βελτίωση των πρωτοβαθμίων ελέγχων είχαμε αυτά τα σεμινάρια που συμμετείχαν πάνω 500 άτομα. Οπότε υπάρχει ενδιαφέρον και από πλευρά κρατών μελών για συμμετοχή, συνεισφορά στην όλη διαδικασία. Οπότε δεν είναι πλέον μόνο δουλειά της Κομισιόν, δεν είναι κάτι το κάνουμε μόνοι μας, αλλά συντονίζονται και τα κράτη-μέλη. Και εκεί πέρα υπάρχει και η δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης. Sur les paiements qui sont, faits à la suite des erreurs, euh, euh, Για τα αχρεωστήτως καταβεβλημένα ποσά που έγιναν αδικαιολόγητα εσείς μπορείτε να τα ξαναπάρετε πίσω διότι τελικά ο φορολογούμενος θα τα πληρώσει δύο φορές δηλαδή αφενός Αυτά τα οποία, το, το καταλάβατε αυτό, δηλαδή αυτά τα οποία ήδη έχει καταβάλει ο φορολογούμενος, Μία Ίσως να ξεκινήσω εγώ και να ζητήσω από πλευρά συναδέλφων να συμπληρωθούν οι πληροφορίες μου. Θα ήθελα να πω φυσικά ότι καθώς γνωρίζετε στο σύστημά μας έχουμε το μέσο, το εργαλείο, τα, μέσα, τα κύρια εργαλεία όσον αφορά για τις επανορθώσεις και αντισταθμίσεις και σίγουρα είναι το πάγωμα αυτό ως μέσο ένα σημαντικό στοιχείο για να εξοικονομηθούν κονδύλια από τον προϋπολογισμό αλλά να έχουμε και ένα κίνητρο για βελτίωση και για τη διαχείριση των ελέγχων και των συστημάτων σχετικών στα κράτη-μέλη. Το 2008 νομίζω ήδη αναφέρθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε τέτοιου είδους ε, χρηματοοικονομικές ε, επανορθώσεις ε, και που απέρεαν και από τους ελέγχους ε, του συνεδρίου και από τους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τέτοιου είδους ε, παρεκκλήσεις ή σφάλματα. Και το να κρίνει κανείς την αποτελεσματικότητα έχει βελτιωθεί αυτή θα έλεγα. Επίσης το 2008 επίσημα παγώσαμε την χρηματοδότηση σε 10 περιπτώσεις που καλύπτουν 31 προγράμματα όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής σχέδια προγράμματα του Ταμείου Συνοχής. Κάνει τη δουλειά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως και τα κράτη-μέλη φυσικά υποχρεούνται να ανακτήσουν τα χρεωστήτως καταβληθέντα στους αποδέκτες που έχουν επωφεληθεί όπου αυτό είναι εφικτό και δυνατό. Όμως έλεγχοι και στοιχεία από τους ελέγχους καταδεικνύουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται αυτό από τα κράτη-μέλη σε περίπτωση και το κάνουν όταν τα σφάλματα οφείλονται στους αποδέκτες που επωφελούνται. Όταν επίσης και τα σφάλματα οφείλονται σε σφάλματα που γίνονται και από την, ε, τις υπηρεσίες της εθνικής διοίκησης, η γραφειοκρατίας και αδυναμίες ε, και του συστήματος ελέγχου αντί να πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται σε σφάλμα τελικού ε, αποδέκτη. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις φυσικά δεν συμβαίνει αυτό. Είναι ο εθνικός προϋπολογισμός όπου επιβαρύνεται με τέτοιου είδους κόστη για την ανάκτηση. Θα έλεγα λοιπόν τούτων λεχθέντων ότι έχουμε στοιχεία σχετικά για αυτά και μπορούν να τα δώσουν ίσως οι συνάδελφοι. Όμως τις δράσεις ε, follow-up μετά από τους ελέγχους και τα αποτελέσματα αυτά ξεκινούν οι διαδικασίες παγώματος πληρωμών ή απέτησης ε, επανόρθωσης. Έχουμε ευελπιστούμε λοιπόν ότι με αυτή τη συνέχεια που θα δοθεί οποιοδήποτε σφάλμα διαπιστώνεται θα μπορέσει να οδηγήσει σε ανάκτηση και θα υπάρχει ανάκτηση. Merci, Madame la Commissaire. Euh, avant une question conclusive, euh, très la simplification. πολύ σύντομα για την απλούστευση. Διαπιστώνοντας το ελεγκτικό συνέδριο ότι μέρος των ελέγχων οφείλεται στην πολυπλοκότητα των ε, κοινοτικών διατάξεων και κανονισμών που μπερδεύουν ακόμη περισσότερα τα κράτη-μέλη επιπροσθέτοντας μέτρα ε, θα, θα, θα, γίνει κάτι, θα προχωρήσετε στην απλούστευση, γιατί και το ελεκτικό συνέδριο και το κοινοβούλιο τη ζητούν. Ναι, προσωπικά πιστεύω και νομίζω ότι ομιλώ εξ ονόματος όλων εκείνων των συναδέλφων και της Επιτροπής που εμπλέκονται στην επιμερισμένη διαχείριση των διαρθρωτικών δράσεων ότι σίγουρα συμφωνούμε για το ότι η απλούστευση μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στο να μειωθούν οι κίνδυνοι σφαλμάτων όσον αφορά τους ίδιους τους αποδέκτες που επωφελούνται από αυτά τα κονδύλια. Επίσης μπορεί και να ανακουφίσει το γραφειοκρατικό βάρος το οποίο υφίστανται και οι αποδέκτες και οι, εθνικοί, ε, και εθνικές διοικήσεις και αρχές. Έτσι λοιπόν, ας το πω έτσι, έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες να προαθούν όλες οι ευκαιρίες απλούστευσης, Απλούστευση αυτών των διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε τέτοιε καταστάσει ότι αυτά τα οποία υποβάλλονται ω κανονισμό από τι Βρυξέλλε επιβαρύνονται και περιπλέκονται περισσότερο στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Και όπω γνωρίζετε για το 2007 και 2013 για αυτή την περίοδο καταβάλαμε προσπάθεια να εισαγάγουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό δράσεων απλούστευση στην χρήση και διαχείριση των διαθετικών ταμείων. Όμω σίγουρα γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει υπάρχει και περαιτέρω δυναμικό. Το Νοέμβριο όταν αποφασίσαμε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξουμε, να εντάξουμε τις δράσεις για την πολιτική συνοχή για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα για την ανάκαμψη και όταν αποφασίστηκαν όλα αυτά προτείναμε επίσης περαιτέρω απλούστευση για το σύστημα και για την χρήση των κονδυλίων των διαθωτικών ταμείων γνωστό αυτό στην Ευρωβουλή γιατί είχα ήδη δύο συζητήσεις με την Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχει προαχθεί αυτή η προσπάθεια από πλευράς του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού όπως διατυπώθηκε, όπως προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο και βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις που εμπλεκόμαστε και όσον αφορά και την Ευρωβουλή και κατά τα τέλη Μαρτίου αν όλα πάνε καλά θα έχουμε μια σοβαρή, ας το πω έτσι, ένα αποτέλεσμα σοβαρό των προσπαθειών απλούστευσης που θα έχουν γίνει πια πραγματικότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά το Περιφερειακό Ταμείο και σε κάποιο βαθμό επίσης και για το Κοινωνικό Ταμείο. Η πρόκληση για μας τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια είναι. Είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και εδώ χρειαζόμαστε και τη βοήθεια της Ευρωβουλής ώστε όλες αυτές οι αλλαγές για την απλούστευση που είναι πάρα πολύ σημαντικέ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ακολουθηθούν από τα κράτη-μέλη που συμμορφωθούν και αυτά και θα υλοποιήσουν αυτή την πολιτική το δυνατόν γοργότερα, ώστε είμαστε πεισμένοι για αυτή την απλούστευση ότι έχει μεγάλη σημασία από πλευρά της. Εκείνο που θέλω να καταστήσω σαφές είναι και συζητείται και από πλευρά ε, συνεδρίου. Οποιαδήποτε απλούστευση θα υπάρξει για τη διαχείριση και το σύστημα ελέγχων δεν πρέπει να υπονομεύει το σύστημα δημοσιονομικών ελέγχων. Αυτό είναι, ας το πω έτσι, κάτι το οποίο πρέπει να μεριμνήσουμε να διασφαλιστεί οπωσδήποτε. Ευχαριστώ άλλες τεχνικές ερωτήσεις. Θα ήθελα να, ρωτήσω, να ζητήσω από την Επίτροπο να μας ε, αναφέρει ποιο είναι το γενικό της αίσθημα, ποια είναι η γενική της εντύπωση, αλλά αυτό μετά από τις ερωτήσεις των συναδέλφων, ο κύριος Ναι, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο. Νομίζω πως φέτος θα είναι πιο εύκολη διαδικασία από την πέρσι. Βεβαίω κατά κάποιο τρόπο είναι δυσκολότερο για μας, γιατί κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που αποφασίσατε μετά από την πίεση του Κοινοβουλίου αποφασίσατε να εφαρμόσετε ξεκίνησαν μόλις το 2008 που σημαίνει βεβαίως πως δεν θα φαίνονται στην διαδικασία απαλλαγής του 2007 ξυπακούεται αυτό Τούτου λεχθέντος. Νομίζω πως κάποια από τα αποτελέσματα που είδαμε όχι μόνο σήμερα αλλά και άλλες φορές είναι πολύ θετικά ιδιαίτερα όσον αφορά τις διορθώσεις και τις αναστολές σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια. Είναι σαφές πως έχουν αλλάξει τα πράγματα και πως πράγματι πολλά από αυτά τα οποία κάνετε έχουν αποτέλεσμα. Τώρα, όπως είπα, είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε σαφή συμπεράσματα. Φαίνεται πως πάμε προς σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί για να περιμένουμε να δούμε τα επόμενα χρόνια πώς θα κυλήσουν τα πράγματα γιατί προφανώς αυτά τα οποία εφαρμόζεται σήμερα θα φανούν ε, σε λίγα χρόνια. Έχω τώρα όμως κάποιες ερωτήσεις για σας. Πρώτα απ' όλα, για τις συμβάσεις αυτές ε, εμπιστοσύνης. Είχατε εντύπωση πως ε, οριστικοποιούνταν αυτές οι συμβάσεις με τις περισσότερες χώρες αλλά τώρα μας είπατε πως είναι μόνο λίγες αυτές οι χώρες μπορείτε να μας ενημερώσετε τι, τι γίνεται σχετικά και άλλη μια ερώτηση για την δυνατότητα να έχουμε προχωρήσει για τον τελικό δικαιούχο από ό,τι μας είπατε σήμερα εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω πως δεν έχετε πλήρη εικόνα και δεν είναι δυνατόν να έχετε πρόσβαση στον τελικό δικαιούχο. Γνωρίζω πόσο μεγάλη πρόκληση είναι αυτό, με τόσα πολλά έργα. Όμως ο δημοσιονομικός κανονισμός ορίζει σαφώς πως θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να έχει αυτές τις πληροφορίες το κοινό πολύ εύκολα. Ναι, αν μπορώ να αναφερθώ σε σχέση με το θέμα του απορρίτου. Ίσως υπήρξε κάποια παρανόηση εδώ, διότι ποτέ δεν είχαμε φτάσει στο να υπογραφεί αυτή η σύμβαση, εμπιστευτική σύμβαση με όλα τα κράτη-μέλη και για να καταστεί σαφές υπογράψαμε την σύμβαση για θέματα εμπιστευτικά, για κάποιες περιπτώσεις επίσης και για το Ταμείο Συνοχής και νομίζω για το συνολικό εγχείρημα βλέποντας κανείς ε, ίσως πολλά περισσότερα θα μπορούσαν να γίνουν. Ναι, η Αυστρία, η, η Ουαλία για την Εσθονία, επίσης Κύπρο και για την η Αγγλία Σε αυτό το επίπεδο βρισκόμαστε, κινούμαστε. Όπως είπα, μόνο για την περίοδο 2000, 2006 ισχύουν αυτά, για αυτή την περίοδο. Για την επόμενη περίοδο έχουμε εντάξει εμ, τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στον κανονισμό ούτως ή άλλως. Αυτό είναι το πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά αυτό το θέμα. Και όσον αφορά θέματα εμπιστοσύνης εμπιστευτικά για τους τελικούς αποδέκτες υπάρχει εδώ μια παρανόηση ίσως με την πρωτοβουλία για την διαφάνεια που ξεκινήσαμε πριν από δύο χρόνια έτσι δεν είναι αν θυμάμαι καλά και για την περίοδο 2007-2013 αυτό που κάναμε τι ήτανε ζητήσαμε από όλα τα κράτη-μέλη να ανοίξουν σε εθνικές ιστοσελίδες τους καταλόγους των τελικών αποδεκτών που εποφελούνται. Και η υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να παράσχει τον κόμβο, το κομβικό σημείο από το, τη δική μας ιστοσελίδα στα εθνικά ιστοδίκτυα και ιστοσελίδες τα εθνικά ε, νομοθετικά πλαίσια είναι διαφορετικά. Ο μόνος τρόπος για να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια ήταν αυτός ο κόμβος, αυτό το κομβικό σημείο. Για τη Γενική Διεύθυνση Regio έχουμε αυτόν τον τομέα που έρχεται σε επαφή κομβικά και με τα κράτη-μέλη και με τις περιφέρειες ε, όπου δημοσιεύονται αυτές οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα, σε αυτόν τον κόμβο. Επίσης προάγουμε και την ε, δυνατότητα πληροφόρησης σε διάφορες δράσεις. Η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών πρέπει να πω δημοσιεύει, δημοσιοποιεί τέτοια στοιχεία τώρα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, υπάρχουν δύο χώρες που δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. Ίσως σήμερα έχει αλλάξει η κατάσταση βέβαια, αλλά πριν από κάποιες μέρες δύο χώρες υπήρχαν και κάποιες περιφέρειες σε ένα κράτος μέλος που δεν είχαν ε, νομίζω ευθυγραμμιστεί. Συνεργαζόμαστε με αυτά τα κράτη για να καλυφθούν αυτά τα κενά στην κάλυψη και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε όλους τους ε, εποφελούμενους αποδέκτες. Αυτά για την περίοδο τώρα 2007-2013. Ευχαριστώ. Για να δώσω κάποια συνέχεια εδώ πέρα, χωρίς να έχω κάποια επιστημονική μελέτη, μου φαίνεται πως η διαφορά στα δεδομένα προς τα οποία μας δίνεται έτσι συνδέσμους μετά είναι πολύ μεγάλη τότε για να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες στο κοινό πρέπει να υπάρχει κάποια τυποποίηση και κάποια δυνατότητα σύγκρισης των δεδομένων από χώρα σε χώρα. Οπότε αν μπορείτε να μας πείτε κάποια λόγια για το πώς σκοπεύετε να το επιτύχετε καθώς αυτό είναι και αίτημα της Επιτροπής αυτής εδώ και χρόνια μάλλον θα έχετε σκεφτεί κάτι και δεν ξέρω εάν μπορείτε μετά γραπτός να μας πείτε ποιες είναι οι χώρες εκείνες που δεν σας έδωσαν ακόμα τις πληροφορίες και τα link που θέλετε. Σας ευχαριστώ. Θα σας τα στείλω αυτά. Να πω το εξής. Σαφώς υπάρχει ο κανονισμός που ορίζει ελάχιστες προδιαγραφές για τα κράτη-μέλη που πρέπει να γίνονται σεβαστές όταν μας δίνουν αυτούς τους καταλόγους των τελικών δικαιούχων. Οι υπηρεσίες εργάζονται τα τελευταία δύο χρόνια και ενθαρρύνουν τα κράτη-μέλη να πάνε πέρα από την ελάχιστη πληροφόρηση. Και ενθαρρύνουμε μέσω των διαπραγματεύσεων την... το να γίνουν έτσι πιο ορατά αυτά τα έργα, η πολιτική να γίνει πιο γνωστή στους πολίτες και αυτό το οποίο βοηθάει βεβαίω στο πλαίσιο αυτό είναι πως ε, για τον κανονισμο 2017 2017-2013 έχει δοθεί περισσότερη έμφαση στα σχέδια επικοινωνίας σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα υπάρχει απέτηση προετοιμασίας της ε, επικοινωνιακής στρατηγικής ε, υπάρχει μια παρουσίαση της δραστηριότητας του έτους οπότε ο συνδυασμός αυτός θα δημιουργήσει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ε, για την πολιτική αυτή από πλευράς του ποιος μπορεί να υποφεληθεί από αυτά και αυτό συνδυασμό με την διαφάνεια, με τη δημοσίευση των καταλόγων δηλαδή από πλευράς κομισιών νομίζω πως εδώ πέρα αυτά θα συνδυαστούν να δώσουν μια κοινή συνισταμένη. Όσον αφορά το ποια περαιτέρω σχέδια θα πρέπει να έχουμε, μπορώ να πω πως η καθημερινή μας δουλειά είναι να ενθαρρυνθεί η καλύτερη ποιότητα των πληροφοριών και σύντομα θα έχουμε την πρώτη αξιολόγηση του που είμαστε και θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα θα δούμε ποια περαιτέρω δράση χρειάζεται, αλλά επειδή υπάρχουν ε, και αυτοί οι υπεύθυνοι επικοινωνιών από το κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και του συναντάμε συχνά στι, Βρυξέλλες, ε, δίνουμε αυτό το, το μήνυμα ότι πρέπει δηλαδή να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες του κανονισμού για τη διαφάνεια. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι να προσθέσουν τίποτα. Απλά και μόνο να υπογραμμίσω αυτά που είπε η Επίτροπος. Η κύρια προσπάθειά μας κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς και για το δεύτερο ήμιση του 2007 ήταν πραγματικά τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες να εντάξουν, να δώσουν αυτά τα αριθμητικά μεγέθη. Μεγάλη προσπάθεια και δαπάνη αναλώθηκε. Δεν έχουμε φτάσει 100% ακόμα. Θα σας γνωστοποιήσουμε σε σχέση με τις περιφέρειες ε, εκείνες που δεν τα έχουν καταφέρει ακόμα, αλλά έχει επιτευχθεί θετική πρόοδος. Τώρα ακολουθεί το δεύτερο βήμα. Πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την καλύτερη χρήση των πληροφοριών που θα είναι διαθέσιμες πλέον. Δύο πράγματα υπάρχουν που πρέπει εδώ να διασφαλίσουμε και να αξιολογήσουμε. Το πρώτο, μπορούμε να κάνουμε κάτι και τι μπορούμε να, θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε τα αριθμητικά μεγέθη να είναι πιο συγκρίσιμα κάπως και πιο διαρθρωμένα, δομημένα στην παρουσίασή τους. Αυτό θα είναι ένα ακαθόδες, δυσχερές θέμα να αντιμετωπιστεί. Πρέπει να δούμε και να το διασφαλίσουμε ότι θα επιτευχθεί. Ένα άλλο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και τα κράτη-μέλη να το πετύχουν προς το συμφέρον τους είναι πέρα από τα αριθμητικά μεγέθη που θα πρέπει να είναι συγκρίσιμα να είναι πιο αναβαθμισμένες οι πληροφορίες ποιοτικά για αυτές που θα παρέχονται για προγράμματα τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους κονδύλια από πλευράς μας. Ευχαριστώ. Για τον κατάλογο έχουμε την κυρία Γκρέσλε, τον κύριο Μούλτερ, την κυρία Γιάλα, τον κύριο Ντιμπλάζιο, Λούτσεβα και την κυρία Κρέλ. Και ολοκληρώνοντας, ε, ναι, άλλοι δύο εδώ, ναι. Παρακαλώ λοιπόν, σύντομα για να είναι δυνατόν. Και συγκεκριμένα, θα σας πω όταν θα έχει λήξει ο χρόνος, η κυρία Γκρέσλε πρώτη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτά που ο Γενικός Γραμματέας μόλις είπε, μπορώ να πω, εσείς οι ίδιοι ε, φταίτε. Γιατί το Κοινοβούλιο είχε συμφωνήσει για μια απλούστευση για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών Υποθέσεων, αλλά η Γενική Διεύθυνση Προπολογισμών, απέρριψε. Η ζωή μα θα ήταν πολύ ευκολότερη αν είχε υιοθετηθεί η πρότασή μα. Αυτά όσον αφορά την υπέρβαση του παρελθόντο, το ξεπέρασμα των προβλημάτων του παρελθόντο. Τώρα, αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα, που είναι καλύτερα και δίνουν ελπίδε για αυτό το, το πεδίο για το μέλλον, ότι θα πάμε καλύτερα. Συνολικά τώρα, απαντήσεις σε, σε σχέση με τις ερωτήσεις ενδιαφέρουσες, γιατί υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τις χώρες. Για πρώτη φορά δίνονται με αυτόν τον τρόπο αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Δεν γνωρίζω εγώ πιο πριν να είχε γίνει κάτι τέτοιο. Θέλω ρητά να ευχαριστήσω γι' αυτό. Η δική μας επιθυμία name and shame, να κατονομάζονται για να ντρέπονται και να ισχύνονται οι υπεύθυνοι. Η Ισπανία πάνω από 50% είναι υπεύθυνη για αυτές τις ε, επανορθώσεις, διορθώσεις των πληρωμών. Πρώτη μου ερώτηση. Ποια ειδικά μέτρα έχετε προβλέψει για την Ισπανία. Έχουμε κι άλλο ένα τέτοιο υποψήφιο που πολλά πράγματα ε, οφείλονται σε αυτόν, στην Ελλάδα δηλαδή, στον τομέα της γεωργίας. Είχε πει σαφώς ε, κάποιες ε, δηλώσεις είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την περίπτωση της Ελλάδας. Τι γίνεται με την Ισπανία, τι υπάρχει σχετικά με αυτήν. Μπορώ να συνεχίσω με τι ερωτήσει μου, ναι. Και θα μπορούσα όπως και ο συνάδελφος Γιώργενσεν, αλλά τέλος πάντων δύο πράγματα τώρα εδώ θα ήθελα να αναφέρω. Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει εκείνοι που προκαλούν τα προβλήματα στα διαθωτικά ταμεία να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους άλλους και μέσα από τους αριθμούς έχουμε την απόδειξη ότι βρίσκεται επικεφαλής η Ισπανία, ακολουθεί η Ιταλία Ξέρω ότι δεν είναι ο τομέας αρμοδιότητάς σας αυτός ε, για το κοινωνικό ταμείο. Έχουμε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο. 90% των σφαλμάτων οφείλονται, τουλάχιστον των διορθώσεων, ε, των οικονομικών διορθώσεων οφείλονται σε αυτές τις τρεις χώρες. Ερώτημα, δεν θα πρέπει να έχουμε ένα ranking όσον αφορά αυτές τις περιπτώσεις ε, και τις διορθώσεις ε, για να επιστήσουμε την προσοχή σε αυτά τα θέματα. Τα κράτη-μέλη υφίστανται τις επιπτώσεις αρνητικά όταν εκείνα τα κράτη που φέρονται σωστά και δεν κάνουν τέτοια πράγματα υφίστανται τις επιπτώσεις για αυτά τα οποία κάνουν άλλοι. Τι γίνεται με την Ισπανία και τι γίνεται με το ranking, την ε, ιεράρχηση, η βαθμολόγηση. Πότε μπορούμε να έχουμε τέτοια στοιχεία βαθμολόγησης. Και μετά και για την προενταξιακή βοήθεια, το μέσο προενταξιακής βοήθειας. Πολλά προβλήματα βλέπουμε να υπάρχουν στην Βουλγαρία, κάπως λιγότερα στη Ρουμανία και οι δύο χώρες ε, τώρα σιγά σιγά αφομοιώνονται, εντάσσονται στα διαθωτικά ταμεία. Ενδιαφέρον θα ήταν να ακούγαμε ποιε προβλέψεις έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι κάνετε δηλαδή εσείς ώστε να εξοπλιστούν οι χώρες αυτές, να είναι σε θέση αυτά τα τεράστια ποσά που τους δίνονται να τα διαχειρίζονται με τον ορθότερο τρόπο και να μην έχουμε μόνο μεγάλα προβλήματα αλλά να μπορούμε να σφίξουμε και τις βίδες για να είναι πιο αποτελεσματικές οι δράσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αλλαγή, πρόταση αλλαγής ε, μεταρρύθμισης ε, του κανονισμού των διαθετικών ταμείων ε, επιτραπέζης. Economic Recovery Plan πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης. Τι γίνεται εδώ και σε σχέση με το ποσοστό σφαλμάτων. Μπορείτε να προβλέψετε τις επιπτώσεις. Ενδιαφέρον θα ήταν να βλέπαμε πού βλέπετε τα δυνατά σημεία αυτού του προγράμματος όσον αφορά ελέγχους και πού βλέπετε αδυναμίες να υπάρχουν όπου θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να το δούμε αυτό. Καλό θα ήταν αν τώρα μπορούσαμε να, να το προσυζητήσουμε για να είμαστε προετοιμασμένοι. Ευχαριστώ. On, Ίσως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τον Νικολάς και μετά με τον κύριο Διευθυντή και να τελειώσουμε. Ναι, για να επανέλθω στο πρώτο ζήτημα που αφορούσε την Ισπανία. Για να σας δώσω κάποιες πληροφορίες για το τι έκανε η Κομισιόν. Μιλώ λοιπόν από τη σκοπιά του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής αναλάβαμε κάποιες δράσεις για να βελτιωθεί η λειτουργία του συστήματος μέσω ενός συστήματος σχεδίου δράσης από τις Ισπανικές Αρχές σε διάφορες περιφέρειες. Έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος, είμαστε ικανοποιημένοι πως σε αρκετές περιφέρειες λειτουργεί επαρκώς το σύστημα, αλλά λόγω αποτυχιών ε, από κάποιους ενδιάμεσους φορείς ελήφθη ε, μια απόφαση αναστολής, ε, θα το δείτε αυτό στον κατάλογο που ελήφθη μια τέτοια απόφαση από την Κομισιόν το Νοέμβριο 2008. Και αυτό επηρεάζει νέα σημαντικούς ενδιάμεσους φορείς. Οι φορείς αυτοί λοιπόν τώρα σύμφωνα με τους όρους αυτής της απόφασης πρέπει να διεξαγάγουν μια σειρά ελέγχων και να μας πούν τι γίνεται με τις παρατυπίες και αν δεν το κάνουν αυτό τότε η Κομισιόν θα περάσει στην επόμενη φάση να εφαρμόσει μια μουσιονομική διόρθωση. Οπότε γνωρίζουμε τις αδυναμίες που υπάρχουν, ε, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα και έχουμε κάποιες διαδικασίες που είτε θα ε, επιφέρουν μια ικανοποιητική βελτίωση ή θα καταλήξουν ε, σε διορθώσει βάρος των Ισπανικών αρχών εάν δεν διορθώσουν αυτό τον κίνδυνο για τον προπολογισμό τη κοινότητα. Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω δύο λόγια για αυτό το παράδειγμα τη Ισπανία, Επιτρέπει την δυνατότητα να φωτίσουμε μέρο των προβλημάτων που καμιά φορά αντιμετωπίζουμε. Τώρα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαμε στην Ισπανία, από τα μεγάλα προβλήματα που είχαμε εκεί και που οδηγεί σε έναν αριθμό συζητήσεων αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Τώρα, αυτό που έγινε στο παρελθόν τι είναι. Οι ισπανικές αρχές είχαν μεταφράσει την οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες στο εθνικό δίκαιο με τρόπο που δεν ήταν 100% ορθός. Όμως μέχρι σχετικά όψιμο χρονικό διάστημα από κανέναν δεν είχαν ενημερωθεί οι Ισπανικές αρχές ότι αυτό δεν έβαινε καλώς και ήταν λάθος και εφάρμοζαν τον Ισπανικό αυτό νόμο, αυτή την Ισπανική ρύθμιση. Εμείς είδαμε, ανακαλύψαμε ότι αυτή η μετάφραση σε εθνικό, μετάθεση σε εθνικό δίκαιο από τους Ισπανούς ήταν λαθασμένη. Το συζητήσαμε και με τους συναδέλφους μας ε, και τα πράγματα τώρα διανοίγονται για να επιληθούν, να επιληθούν αυτά τα ζητήματα. Το θέμα είναι με το παρελθόν. Πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα όταν ε, ένας λανθασμένος εθνικός νόμος σωστά εφαρμόστηκε. Τα λέω όλα αυτά για να επιστήσω την προσοχή ότι με την περίπτωση naming and shaming να ονοματίσουμε κάποιους για να κατηγορηθούν και να εσχυνθούν δεν είναι η σωστότερη ακριβώς περίπτωση εδώ καμιά φορά. Ίσως να πω και δύο λόγια για τη Βουλγαρία και την Ρουμανία στη συνέχεια. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να αναφέρω το εξής. Στην περίπτωση της Ρουμανίας, καθώς αφορώνται τα διαθωτικά ταμεία και ιδιαίτερα το Περιφερειακό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, πρέπει να πω ότι η συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές βαίνει καλός. Δεν έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχουν μείζωνα προβλήματα σχετικά μέχρι σήμερα. Όμως πρέπει να προσθέσω όσον αφορά την περίοδο 2007-2013 ότι βρισκόμαστε ακριβώς στην πρώτη φάση, πρώιμη στιγμή αυτή ακόμα για να συναγάγουμε συμπεράσματα. Τώρα στην περίπτωση της Βουλγαρίας τι γίνεται. Θα έλεγα σχετικά και μας εκπλήσει αυτό ότι μάλιστα ακόμα και για τη Βουλγαρία η πολιτική αυτή ως προσέγγιση ως ε, παράδειγμα λειτουργεί καλά. Και σε σχέση με το παράδειγμα που είχαμε, σε αυτό αναφέρομαι, για την χρηματοδότηση οδικού δικτύου οδών ε, και για τη διαφθορά σε σχέση με τη Βουλγαρία. Μετά από 24 ώρες ε, συνειδητοποιήθηκε αυτό το πρόβλημα από πλευράς μας. Είχαμε ήδη συμφωνήσει με τους Βουλγάρους συναδέλφους εταίρους ότι θα πάγωναν οι πληρωμές, ότι δεν θα ήταν δυνατόν να καταβληθούν τέτοιες πληρωμές, θα διεκόπεται η ροή χρηματοδότησης και όταν θα βλέπαμε ότι αυτό θα ήταν ένα πιο μακροπρόθεσμης πνοής ε, πρόγραμμα από ό,τι στην αρχή, επίσημα ακολουθήθηκε μια διαδικασία παγώματος ε, και τώρα σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς μας τώρα περιμένουμε να επιληθεί ικανοποιητικά από τη βουλγαρική πλευρά αυτό το πρόβλημα παρέχοντας όποια υποστήριξη μπορούμε στους ε, αρρωγείς τους Βουλγάρους εκείνοι όμως είναι υπεύθυνοι για την επίλυση αυτού του πρόβλημα προβλήματος. Όταν θα έχει επιληθεί αυτό το πρόβλημα με δειγματοληπτικούς ελέγχους επιτόπου και διασφαλιστεί ότι έχει αντιμετωπιστεί, θα ξανανοίξουν οι στρόφιγγες για χρηματοδότηση και θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση. Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι όταν είναι προφανές ότι υπάρχει κάπου ένα πρόβλημα, το σύστημα γοργά και συστηματικά όταν εφαρμόζεται όπως πρέπει, έχει αποτελέσματα όπως τώρα. Και έτσι φαίνεται ότι λειτουργούν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν υφίστανται προβλήματα. Αυτό σημαίνει απλά ότι με τη βάση της λειτουργίας του συστήματος μέχρι σήμερα καθώς μπορούμε να κρίνουμε έχουμε αποκομίσει την εντύπωση ότι ναι μάλιστα μπορούμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αυτό το σύστημα, με αυτόν τον τρόπο. Όποτε θα διαπιστώνεται και θα υπάρχει πρόβλημα θα παγώνουν οι πληρωμές. Και αυτό φυσικά πιέζει και οθεί τα κράτη-μέλη, είναι ένα κίνητρο για να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν τα προβλήματα. Και πρέπει να πω ότι μεγάλες προσπάθειες καταβάλλονται ή καταβλήθηκαν από τη Βουλγαρία, στη Βουλγαρία για να συμμορφωθούν και να προχωρήσουν έτσι. Θα δούμε λοιπόν δειγματοληπτικά με ελέγχου αν αυτό έγινε, αν αυτό επαρκεί και έτσι θα συνεχίσουν. Σύντομα να πω κάποια πράγματα για το ποσοστό σφάλματος στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης γιατί και αυτό τράβηξε την προσοχή μας. Όπως είπα, θεωρώ πως η απλοποίηση εν γίνει σωστά μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα στη μείωση του ποσοστού σφάλματος, γιατί οι απλούστεροι κανόνες ε, εφαρμόζονται και πιο εύκολα και είναι πιο ευνόητοι. Οπότε αν καταφέρουμε να εξηγήσουμε τώρα στη δουλειά μας με τα κράτη-μέλη και τις εχειριστικές αρχές πώς θα χρησιμοποιηθεί οπλοποιημένος κανονισμός, μπορούμε να συνεισφέρουμε στη μείωση του ποσοστού σφάλματος. Γνωρίζουμε όμως πως ε, ε, κάποια απλοποίηση μπορεί επίσης ε, να οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού σφάλματος εάν δεν γίνει σωστά. Γι' αυτό έχουμε επαφές και με το ελεγκτικό συνέδριο να δούμε πως υπάρχουν κάποιες απόψεις ε, ειδικών από εκεί για να δούμε πού πιθανώς είναι ο κίνδυνος. Αλλά παραδείγματος χάρη να αυξήσαμε την πρόσβαση στην τεχνική αρρωγή μέσω του γραφείου του προγράμματος Jaspers, αυξήσαμε τις δυνατότητες του συστήματος για την προετοιμασία των μεγάλων έργων όπου είναι υψηλότερος ο κίνδυνος Οπότε προτείνουμε αυτή τη δράση που θα μας βοηθήσει να μειώσουμε το ποσοστό σφάλματος σε αυτό το τομέα. Επιπλέον βεβαίως όταν ε, ο κανονισμός ε, περάσει την διαδικασία την ε, νομοθετική θα εκδώσουμε και κάποιες καθυστήριες γραμμές. Το συζητάμε ήδη με την Κόκοφ, έχουμε κάποιες συναντήσεις για να δούμε πού μπορεί να υπάρχει κίνδυνος κατά την εφαρμογή των απλοποιημένων κανόνων. Να πω επίσης πως η όλη αυτή η διαδικασία γίνεται ξεκινώντας από την υπόθεση ε, εργασίας πως δεν ε, υπονομεύει το σύστημα ελέγχου και δεν δημιουργεί νέους κινδύνους στον έλεγχο του προπολογισμού. Και αυτό οφείλουμε να διαπιστώσουμε. Τώρα για τον πίνακα κατάταξης αυτών που παραβιάζουν, που δεν έχουν αποτελέσματα και συνεισφέρουν στο ποσοστό σφαλμάτων στην εφαρμογή. Πράγματι δεν έχουμε κάποιον κατάλογο των κρατών μελών, αλλά είναι γνωστές οι πληροφορίες Οπότε νομίζω πως όλοι ξέρουν που είναι τα λάθη. Και επιπλέον, όταν ε, αποφασίζουμε τη στρατηγική ελέγχου, με βάση τις εμπειρίες ε, μεμονωμένων κρατών μελών, γνωρίζουμε που είναι υψηλότερος κίνδυνος και το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη. Οπότε θεωρώ πως εμείς ε, στην Κομισιόν και τα κρατημέλη έχουμε επαρκείς πληροφορίες για το πού είναι συχνότερα τα προβλήματα και οφείλω να πω πως ε, δεν είχαμε σκεφτεί ποτέ να συντάξουμε ένα τέτοιο κατάλογο. Οπότε... Θα θέλαμε μια τέτοια, ένα τέτοιο κατάλογο βαθμολόγησης. Έχω την εντύπωση ότι έχει νόημα να είμαστε προσεκτικοί στις πληρωμές. Αυτές μπορεί κανείς ε, πιο γρήγορα να τις σταματήσει από ότι να ζητήσει να ανακτήσει εκ των υστέρων κάποια ποσά. Και γι' αυτό τα οποία είπε ο Γενικός Διευθυντής για τη Βουλγαρία φαίνεται ότι αυτό υπογραμμίζεται. Ο κύριος Μούλτερ ζήτησε τον λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω επενώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μεγάλη προθυμία να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις από την Ευρωβουλή διαπιστώνεται. Δεν δίνεται εντύπωση ότι κάτι αποκρύπτεται, αυτό είναι, θέλουν να αποκρύψουν κάτι, αυτό είναι κάτι θετικό. Είναι όμως πραγματικά πολύ βραδύς ο αριθμός που ακολουθείται για την επίτευξη πρόοδου και αν δει κανείς σε σχέση με την έκδοση μιας θετικής δήλωσης, θετικής DAS, έχουμε ένα 11% το οποίο διαπιστώνεται και έχουμε μεγάλη οδό, μεγάλη πορεία να καλύψουμε. Έχει πολλή δουλειά να γίνει για τη χωρίς απαλλαγή. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το πρόγραμμα δράσης έχει στεφθεί με επιτυχία. Είναι δεν ξέρω αν 37 ε, μέτρα έχουν πλήρως υιοθετηθεί, αλλά για το πρόγραμμα δράσης, όπως λένε σύμφωνα με αυτούς, ήταν σε μεγάλο βαθμό επιτυχές. Αν συμβαίνουν όλα αυτά, Πώς αυτό δεν αντανακλάται στα στοιχεία. Ποια είναι η επεξήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι μπορούν να πούν, πώς μπορούν να πούν ε, σήμερα αυτό το απόγευμα ότι ήταν επιτυχές το πρόγραμμα δράσης και να έχουμε τέτοια μεγέθη που αποκαλύπτονται εδώ. Θέλω να επανέλθω τώρα στη διαδικασία για το 2009. Είχα ε, την ιδέα και υποστηρίχθηκε ότι 12% των κονδυλίων του ε, Διαθωτικού Ταμείου θα έπρεπε να εγγραφεί σε αποθεματικό και θα μπορούσε μεταξύ πρώτης και δεύτερης ανάγνωσης να προσεγγίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη και να απαντηθούν στις ερωτήσεις και παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να μπορεί περισσότερα να δίνονται από τα κράτη-μέλη από ό,τι στις ανακεφαλαιώσεις ε, των κρατών μελών. Καλό θα ήταν 12% να εγγραφεί στο αποθεματικό μεταξύ πρώτης και δεύτερης ανάγνωσης. Αυτό θα επικέντρωνε τα κράτη-μέλη και θα τα πίεζε πολύ περισσότερο και θα μπορούσε να είχε βοηθήσει και την Επιτροπή περισσότερο. Κατανόησα ότι ήταν εναντίον ε, αυτή τη προσέγγιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να επιβεβαιώσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν ναι, αν γίνεται αυτό τότε γιατί συμβαίνει αυτό. Σε τι οφείλεται. Διότι νομίζω πολύ πιο εύκολο θα ήταν να είχαμε τις σωστές δομές διασφαλισμένες προτού αναλυφθεί δράση. Αν δεν υπάρχουν τέτοιες δομές μπορεί κανείς να είναι υπερήφανος για την ανάκτηση ενός ενάμιση δις μεγάλα ποσά αυτά. Όμως το γραφειοκρατικό κράτο, κόστος το οποίο ε, μπλέκεται εδώ και συνεπάγεται μια τέτοια δράση θα μπορούσε να είχε αποφευθεί. Θα μπορούσαμε να είχαμε βοηθήσει, να είχε υπάρξει βοήθεια για να είχε επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Δεν υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή Προπολογισμών η ιδέα αυτή τη Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Και έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε σε αυτήν την κατάσταση. Όμω παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα βοηθούσε αν ευθύ εξ αρχή μπορούσαμε να εγγράφαμε κάτι στο αποθεματικό θα σας βοηθούσε εσάς με τον καλύτερο τρόπο να αναγκάσετε τα κράτη-μέλη να συμμορφώνονται με τα όσα εσείς απαιτείτε. Και δύο, ε, ένα, μια τελευταίο σχόλιο για τη Βουλγαρία και Ρουμανία. Πρέπει να πω ότι υπερψήφισα εγώ για την διεύρυνση στο παρελθόν και ήμουν πάντα στεναρός υπέρμαχο και υποστηρικτή τη διεύρυνσης και για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία διότι πιστεύω ότι η διεύρυνση διασφαλίζει και ενδυναμώνει την δημοκρατία πανευρωπαϊκά. Δεν χρειάζεται εμένα λοιπόν να με πείσετε ότι είναι κάτι το θετικό η διεύρυνση τα γεγονότα, τα στοιχεία μιλάνε όμως και εδώ δείχνουν ότι υπάρχουν, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα εκεί. Ίσως ε, ήταν ε, θέμα να απευθυνθεί και ερώτηση στον Όλυ Ρεν. Πώς μπορεί να επεξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δίνονται διασφαλίσεις στην Ευρωβουλή και υπήρξε και η πίστη ότι όλοι οι μηχανισμοί μπορούσαν να λειτουργήσουν, μηχανισμοί ελέγχου και μετά αποκαλύπτεται ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε και είχαμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Ευχαριστώ. Uh, ναι όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ε, και εγώ προέρχομαι από νέο κράτος μέλος όπως το λέμε. Όπως ξέρετε έχουμε και στην προενταξιακή περίοδο αυτά τα ταμεία για να προετοιμάσουμε τις υποψήφιες χώρες για τη συμμετοχή τους στην πολιτική. και ειδικά το ΙΣΠΑ ήταν πάντα ένα τέτοιο μέσο και έχουμε τώρα τον ίδιο μηχανισμό με το μέσο το πρενταξιακό που με κάτι παρόμοιο αυτό το οποίο έχουμε στα διαρθρωτικά ταμεία. Οπότε στην προενταξιακή περίοδο έχουμε και τις διαπραγματεύσει για το να στηθούν συστήματα καλής ποιότητας και υπάρχει και μία περίοδο, μια περιοδο μια εξάσκησης ε, μέσω των μέσων ΙΣΠΑ και ΙΠΑ. Βεβαίω πρέπει να λάβουμε υπόψη πως ε, αυτές είναι πολιτικές που συχνά είναι ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος για την αποτελεσματικότητα λειτουργίας πολλών άλλων συστημάτων ε, και του και της δικαιοσύνη και του δημοσιονομικού τομέα, π.χ. οτιδήποτε αφορά τις δημόσιες προμήθειες στην εσωτερική αγορά. Οπότε το βάρος εδώ πέρα είναι και ο πρακτικός έλεγχος της συμμόρφωσης των εθνικών συστημάτων σε πολλούς τομείς συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Γι' αυτό μέσω αυτής της πολιτικής ανακαλύπτουμε όλη αυτή την αναποτελεσματική λειτουργία. Πριν υπάρξει καν ένταξη θα έλεγα πως σε πολλές περιπτώσεις βεβαίω, δεν το υπερασπίζομαι γιατί ξέρω πως πρέπει να διασφαλίσουμε ε, πλήρη διασφάλιση πριν από την ένταξη αλλά η πιθανότητα το σύστημα να φαίνεται σωστό και να εκπληρώνει όλα τα κριτήρια στα χαρτιά μετά στη λειτουργία του να μην λειτουργεί αποτελεσματικά. Π.χ. οι νόμοι για τις δημόσιε προμήθειε. έχουμε δει πολλές περιπτώσεις, οποίες έχουμε έναν εθνικό νόμο που συμμορφώνεται πλήρω με το κοινοτικό δίκαιο, αλλά μετά οι εφαρμοστικοί κανόνες είναι τόσο πολύπλοκοι που καταλήγουμε σε επιχειρήσεις που δεν χρησιμοποιούν αυτό το, το σύστημα και δεν, ε, δεν λειτουργούν οι νόμοι τελικά και παραπιάζουν το κοινοτικό δίκαιο αυτή την κατάσταση. Και οι άνθρωποι από το ΕΚΤ ε, και από αλλού που εργάζονται επί τόπου ανακαλύπτουν παρατυπίες στα συστήματα που στα χαρτιά φαίνεται ότι συμφωνούν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο αλλά οπωσδήποτε τα συμπεράσματα από την ένταξη Βουλγαρίας και Ρουμανίας πρέπει να βγουν και είμαι σίγουρο, ε, σίγουρη πως αυτή τη στιγμή η Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης τα εξετάζει αυτά και εξετάζει τις πτυχές των συστημάτων με κάπως διαφορετικό τρόπο από το παρελθόν. Είμαι σίγουρο πως αυτό ακριβώς συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά όπως είπε και ο κύριος ε, Γενικός Διευθυντής, ποτέ δεν είναι αργά, γι' αυτό συνεργαζόμαστε με αρχές, κάνουμε τους ελέγχους των συστημάτων, χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να μην υπάρχουν παρατυπίες ε, στην εκταμείευση των ε, χρημάτων, αλλά υπάρχει αυτή η πρόκληση να δούμε πώς θα έχουμε μεγαλύτερη διασφάλιση πριν από την ένταξη ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Όσον αφορά το σχέδιο δράσης, και το πότε θα έχει αποτελέσματα. Έχουμε αρκετές ε, πρωτοβουλίες που σχετίζονται και με το κλείσιμο της περίοδου 2000-2006. Οπότε ελπίζουμε πως το κλείσιμο θα μας δώσει δυνατότητα να αποδείξουμε πως ε, το ποσοστό σφάλματος θα είναι ήδη χαμηλότερο και θεωρώ πως ε, το 2010 όταν θα έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία θα μπορέσουμε να κάνουμε μια εκτίμηση προς την αρχή του προϋπολογισμού για να δείξουμε πως ε, το ποσοστό σφάλματος που απομένει για τα προγράμματα 2000-2006 ε, να δούμε ποιο θα είναι αυτό και αυτή θα είναι η στιγμή που και εμείς θα πρέπει να αποδείξουμε πως οι δράσεις οι οποίες έχουμε ε, λάβει έχουν και αποτέλεσμα. Επίσης και μέσω των επανορθωτικών πράξεων που κάνουμε τελευταία χρόνια, μέσω των διορθώσεων που αναφέραμε, για αυτά τα οποία ενημέρωσε και ο Διευθυντής, όλα αυτά ξεσκαρτάρουν και τις ε, δαπάνες της ε, αντικανονικές, οπότε μιλήσαμε επίσης και για σημαντική πτώση του, του σφάλματος στις ενδιάμεσες πληρωμές 2007-2013, οπότε χωρίς να είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη, ρεαλιστικά θα έλεγα πως ε, θα πρέπει να αρχίσουμε να, να έχουμε αποτελέσματα για τον κύριο όγκο των δαπανών του χρόνου οπωσδήποτε. Αυτή είναι η κρίση μου, αλλά πιστεύω πως και η συζήτηση και το γεγονός ότι είχαμε το σχέδιο δράσης, είχαμε αυτή τη δύσκολη συζήτηση για τα συστήματα των κρατών μελών και τους μηχανισμούς ε, ήδη έχει οδηγήσει σε ευαισθητοποίηση των κρατών μελών εντός των συστημάτων διαχείρισης κάτι το οποίο οδηγεί σε μείωση του ποσοστού Σε σχέση με αυτό το οποία κάνει απευθείας η Κομισιόν. Για τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν Πρέπει να προχωρήσουμε λίγο κύριε Επίτροπε. Πρέπει να δούμε και το ρολόι. Κυρία Αγιάλα έχει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κρίμα που η της ε, έφυγε αλλά ε, έφυγε για λόγους ανωτέρας βίας πάντως ε, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μπρί για το εξαιρετικό του ερωτηματολόγιο και να τον ευχαριστήσω και για την συμβολή του στην επίλυση όλης αυτής της επίπονης διαδικασίας που είναι η απαλλαγή. ο συνάδελφος έψαξε να βρει την ρίζα του προβλήματος των λογαριασμών που δημιουργούν πονοκεφάλους ε, στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη και η Κομισιόν επίσης βοήθησε να αποφύγουμε κινδύνους. Και φαντάζομαι ότι η Ισπανική κυβέρνηση βρίσκεται στη διάθεση της Κομισιόν για οποιαδήποτε πληροφορία. Τώρα για την Επίτροπο. Σε αυτή τη φάση της οικονομικής κρίσης, σε ποιο βαθμό η εφαρμογή του σχεδίου δράσης και στις πιο σημαντικές του πλευρές, δηλαδή την απλούστευση που διευκολύνει τη δράση και τον έλεγχο, πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με την ευκαιρία δηλαδή και της κρίσης για να βελτιώσουμε αυτήν την διαδικασία απλούστευσης ε, το θέμα των ε, αχρεωστήτως καταβληθέντων πληρωμών, την ίσπραξή τους μετά κλπ. Πώς μπορούμε λοιπόν να ενισχύσουμε τον, το, το σύστημα των ελέγχων σε αυτή τη φάση είναι η καλή στιγμή για το θέμα τώρα που έθεσε ο Γενικός Διευθυντής ε, για την ποιότητα, μα όλοι περιμένουμε αυτή την ποιοτική αναβάθμιση. Εγώ θεωρώ ότι όλη η διαδικασία βελτιώνει ιδιαίτερα την δυνατότητα των κρατών μελών να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο το, έστω και το ένα ευρώ του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Εμείς ε, Θέλουμε να δικαιολογήσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ, αλλά από την άλλη μεριά θέλουμε και να δικαιολογήσουμε ότι όλα τα ευρώ μέχρι και το τελευταίο ευρώ που ξοδεύτηκε, ξοδεύτηκε σωστά. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω, να ζητήσω από τον κύριο Όντι, Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Ντί, ευχαριστώ και την Κομισιόν και τα λοιπά. Θέλω να ζητήσω το πώς μπορούμε να καταλήξουμε στον ελαχιστότερο των κινδύνων. Πώς προσεγγίνουμε λοιπόν σε αυτό. Και μετά Θα ήθελα να συζητήσουμε και το θέμα της μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί το ελεγκτικό συνέδριο. Βέβαια αυτή η συζήτηση θα γίνει στην επόμενη στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Διότι με το ελεγκτικό συνέδριο όσο δεν έχουμε καθαρά τα πράγματα είναι σαν να έχουμε μια δαμόκλειο σπάθη στο κεφάλι μας. Και όπως λέει και η κυρία Ντανούμπερ σχετικά με τους πραγματικούς κινδύνους. Θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται οι έλεγχοι ως κάτι το ευχάριστο. Θα έπρεπε να θεωρείται ο κάθε έλεγχος ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε. Κυρία Γκρέσλερ, χώρες όπως η Ισπανία και η Γερμανία διότι ναι μεν η Ισπανία στον κατάλογο αλλά και η Γερμανία δεν υπέγραψε αυτό τον κατάλογο εμπιστοσύνης. Τέλος πάντων για αυτά τα συμβόλαια πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο ελέγχου ή όχι. Παρακαλούμε τώρα μια συντομότερη απάντηση από την ερώτηση. Δεν ήταν ερώτηση, αλλά σε σχέση με την Ισπανία αυτό που μπορώ να πω είναι ότι από ό,τι γνωρίζω είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το σύστημα και γι' αυτό το να υπογραφεί μια σύμβαση εμπιστευτική θα απαιτούσε μια ειδική συμφωνία μεταξύ του εθνικού και του περιφερειακού αυτού ε, πλαισίου. Ίσως ένας από αυτούς είναι ένας από αυτούς τους λόγους για τους οποίους δεν μπόρεσε η Ισπανία να υπογράψει μια τέτοια σύμβαση εμπιστευτική, εμπιστοσύνης. Αλλά για την Ισπανία ε, είναι ένα από τα κράτη-μέλη που ομολογεί, αναγνωρίζει τα σφάλματα και ξεκινά τη διαδικασία, ας το πω έτσι, εκαθάρισης των κακώς εχόντων. Είναι ένας πολύ έντιμος εταίρος μέσα σε αυτό σε αυτή την προσπάθεια, στην προσπάθεια αντιμετώπισης ε, των μολυσμένων, ας το πω έτσι, προγραμμάτων που πρέπει να εξηγιανθούν. Πρόεδρος, είναι σημαντική αυτή η επισήμανση και αλλού πρέπει να ακολουθείτε. Προσπάθεια προστασίας ε, των ε, οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ε, εκείνοι που έχουν τα περισσότερα σφάλματα δεν είναι οι μεγαλύτεροι απαταιώνες. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και πρέπει εδώ να διαφοροποιούμαστε σε σχέση με αυτά από πλευρά εισηγητού. Ο κύριος Δεμπλάζιο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αφού άκουσα όλες τις παρεμβάσεις που έγιναν, έχω πλέον την εντύπωση πρέπει να πω ότι η λειτουργία και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών που ακολουθήθηκε, παρόλα αυτά ο ασθενής παραμένει θανάσιμα άρρωστος και υπάρχει ο κίνδυνος να πεθάνει στα χέρια μας. Παρόλα αυτά θέλω στην Επιτροπή και ιδιαίτερα στην, προς την Επίτροπο να ευχαριστήσω, να εκφράσω ευχαριστίες για το ότι προσπάθησε τουλάχιστον με βάση τις προτάσεις μας να υιοθετήσει νέα μέτρα. Και ελπίζω ότι σύντομα, γοργά, θα ακολουθήσουν επιτυχίες. Παρόλα όσα τώρα διαπιστώνει το ελεγκτικό συνέδριο, ήδη βρισκόμαστε στον κίτρινο τομέα όσον αφορά τα περισσότερα κράτη-μέλη. Και παρόλα αυτά, πρέπει να πω, παρόλα αυτά, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ακόμα. Υπάρχουν ε, πολλές ε, πληρωμές που έγιναν που δεν ε, έγιναν σωστά. Ας μιλήσουμε για την Ουγγαρία, για την πατρίδα μου δεν είναι απλά τα πράγματα. Η πρόσβαση στα κονδύλια δεν απλουστεύθηκε. δεν διευκολύνθηκε. Στην, ε, στις Βρυξέλλες δακτυλοδείχνουν ως υπέτειους, ως ένοχους τους Ούγγρους. Εμείς ε, δακτυλοδείχνουμε τους ε, ε, κοινοτικούς υπαλλήλους στις Βρυξέλλες ως υπεύθυνους. Τα πράγματα δεν έχουν βελτιωθεί λοιπόν. Η ερώτησή μου, πώς είναι δυνατόν να έχουμε 11%. Πώς καταλήξαμε σε αυτό το 11%. Υπήρξε είναι ένα σύνολο που καλύπτει όλα τα προηγούμενα συμβάντα ή ισχύει μόνο για αυτό το τρέχον έτος. Αν συμβαίνει αυτό, αν ισχύει μόνο για το τρέχον έτος, τότε δεν θα μπορούμε να υπολογίζουμε ότι θα υπάρξουν βελτιώσεις. Δεν βελτιώνονται τα πράγματα. 3,5 δις ευρώ έχουμε. 3,5 δις ευρώ επαναλαμβάνω που υπό τους ελέγχους αυτούς ε, καταδεικνύουν ε, ανομαλίες και παρατυπίες. Πώς μπορούν να ανακτηθούν τέτοιου ύψους κονδύλια. Και όσον αφορά την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, το ελεγκτικό συνέδριο έχει τους μηχανισμούς ε, αυτούς που επένεσε και ότι είναι λέει καλύτεροι από ό,τι στο παρελθόν. Όμως από αυτό εγώ συνάγω ότι το πρόβλημα ούτε καν στο επίπεδο των κρατών μελών δεν είναι αλλά είναι στο επίπεδο των τελικών χρηστών ή καταναλωτών ας το πω έτσι διότι τα περισσότερα σφάλματα προέρχονται ή οφείλονται στις ε, κρατικές ας το πω έτσι διαδικασίες ε, κύρωσης ε, ή προμήθειας και δείχνει αυτό ότι κάτι από πλευράς παρατυπιών οφείλεται στις, ε, στους τελικούς χρήστες. Επανέρχομαι στην Ισπανία. Στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, για όποιον διάβασε προσεκτικά την έκθεση, αναφέρεται ότι παράλληλα με αυτά τα μεγάλα προβλήματα υπάρχουν και άλλα προβλήματα που αναφύονται εντωμεταξύ, που παρουσιάζονται και στην ομοθεσία, στην ομολογία για παράδειγμα. Κάποια σφάλματα τα οποία θεωρούμε σφάλματα, τα κράτη-μέλη δεν τα θεωρούν σφάλμα, δεν τα θεωρούν λανθασμένα. Και αν αυτό συμβαίνει, αν οι ορισμοί δεν είναι συγκρίσιμοι και δεν είναι ίδιοι, αν θέλουμε να συγκρίνουμε αχλάδια με μήλα, δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σωστά συμπεράσματα. Όμως ερώτηση προς το Συμβούλιο, τώρα θέλει να παρέμβει, προς το ελεκτικό συνέδριο με συγχωρείτε, θέλετε να παρέμβετε εσείς ε, κυρία για το 11% και το τι συνεπάγεται αυτό. Thank you. Μάλιστα, ευχαριστώ. Η ερώτηση αφορά τους τύπους σφαλμάτων που υπάρχουν και αν έγιναν αυτά τα σφάλματα κατά το έτος που συζητάμε, το 2007 ή όχι και για τις ε, επιστροφές που ζητήθηκε να ε, γίνουν ε, σε σχέση με το 2007 και για το σύνολο της περίοδου 2000-2007 το σφάλμα αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι υπήρξε υπερβολικός υπολογισμός του κόστους και πρέπει να υπάρξει ανάκτηση. Μπορεί να είναι σφάλμα υπολογισμού, μπορεί να είναι σφάλμα εκπαραδρομής, μπορεί να είναι συνδυασμός και των δύο. Επιλεξιμότητα σφάλμα σημαίνει ότι δεν είναι σύμβατη η επιστροφή, η ανάκτηση με τους κανονισμούς. Σφάλμα εκ παραδρομής γίνεται όταν συμπεριλαμβάνεται ένα κόστος το οποίο δεν έχει, δεν έχει δαπανηθεί ή και δεν υπάρχουν ε, αποδείξεις γι' αυτό και για, την, ε, για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Ίσως εδώ μπορεί να υπάρξουν σφάλματα συμμόρφωσης ε, και εδώ να υπάρχει το πρόβλημα το οποίο εκ παραδρομής παρουσιάζεται και σε σχέση με το ποσοστό σφάλματος το οποίο υπολογίζει το ελεγκτικό συνέδριο και στα ποσοστοποιήσιμα και στα μη ε, υπολογίσιμα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα σφάλμα κοινό και συχνό. Επίσης ο λανθασμένο, λανθασμένος υπολογισμός όσον αφορά τίτλους, κατηγορίες, πράγματι αυτά αφορούν το 2007. Θα ήθελα να πω δίνουμε αξία όσον αφορά την ε, υποστήριξη. Πρέπει να πούμε ότι η ετήσια έκθεση του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιμετωπίζει, αναφέρει αυτό το πρόβλημα. Το, ο συνολικός όγκος ήταν μεγαλύτερος και εντάσσουμε αυτό ως εν μέρη αποτελεσματικό. Τώρα, αν αυτό είναι μεγάλη πρόταση, ή όχι, αυτό είναι θέμα που θα πρέπει η Ευρωβουλή να αξιολογήσει. Εμείς όμως θεωρούμε ότι μερικά αποτελεσματικά ήταν τα πράγματα. Δεν έχουμε όμως ακόμα αντιμετωπίσει το ποσοστό σφάλματος όπως θα έπρεπε. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Οι περισσότερες εξηγήσει δόθηκαν από την κυρία Κόγιο Λάιτ. Τώρα το πρόβλημα του 11% το οποίο αναφέρεται στις πληρωμές για το 2007 και η συνάρτηση με το πρόγραμμα δράσης ε, που υιοθετείται και εφαρμόζεται. Με κάθε σαφήνεια όταν ξεκίνησε το 2008 το πρόγραμμα δράσης οι έλεγχοι για τις δαπάνες του 2007 ευρισκόντουσαν υπό εξέλιξη καθοδόν ήδη. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι σημειώνεται δεν υπάρχει κάποια αλλαγή για το 2007 πρώτον. Προς έκπληξη όχι. Μια και ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προηγούμενα μπορεί να είμαι πολύ σύντομος. Μπορώ να είμαι πολύ σύντομος. Γίνεται η προσπάθεια να προωθήσουμε, να προαγάγουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν το δικό τους ελεκτικό έδρο, έργο μέσω των ε, <clears throat> μέτρων που υιοθετούνται. Για το αποτέλεσμα αναμένουμε όπως την, κατά την περίοδο 2000-2006 κατά την καταληκτική περίοδο του προγράμματος και για την περίοδο 2007-2013 θα μπορούμε να κρίνουμε όταν θα έχουμε τις ε, πραγματικές ενδιάμεσες δαπάνες για αυτή την περίοδο. Και στις δύο περιπτώσεις 2010-2011 ε, θα έχουμε τέτοιου είδους αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούτσεβα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, κύριε και κύριοι. και εκπρόσωποι του ελεκτικού συνεδρίου. Είναι μια ευκαιρία αυτή που έχουμε να σχολιάσουμε προβλήματα τα οποία συναρτώνται με την αποτελεσματική χρήση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη-μέλη και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες επίσης. Πρέπει να προβληματιστούμε για μέτρα για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Τα στοιχεία στην έκθεση και στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι υπάρχει μια κάποια βελτίωση στη διαχείριση των, της καταβολής κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρότι το ποσοστό σφάλματος είναι 18% λέει ο ομιλήτρια. Κάνοντας λόγο για σφάλματα, παρατυπίες και τέτοιου είδους λάθη θα ήθελα να διατυπώσω κάποιες ερωτήσεις. Ίσως σε σχέση με τις παλαιότερες ε, χώρες μέλη που έχουν μεγαλύτερη πείρα μπορούν να δείξουν πώς επαναλαμβάνονται αυτά τα σφάλματα και με ποιο τρόπο και με ποιο τρόπο μπορούμε να παρα, κολλήσουμε να αποφύγουμε τέτοιου είδους σφάλματα, να μην υπάρχει δηλαδή διαρκώ το ίδιο σφάλμα το οποίο θα γίνεται και ευθύ εξ αρχή να βοηθήσουμε να μην γίνεται αυτό ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές. κανοντά λόγο για το Ταμείο ε, ε, προετοιμασία για την Ένταξη που ε, μας αφορά, νομίζω σε μια περίοδο προένταξης πραγματικά παίρνουν τέτοιου είδους χώρες σημαντική αρρωγή, σημαντικά κονδύλια που τους υποστηρίζουν από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προετοιμαστούν για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια αυτή πρέπει να είναι σεβαστές διάφορες ε, ε, προθεσμίες, ε, όροι, προϋποθέσεις. Νομίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όλα τα αναγκαία μέτρα και για έλεγχο υιοθετήθηκαν και λειτουργήσαν κατά τη διάρκεια της προενταξιακής περίοδου ώστε να μην ε, υπήρχαν προβλήματα, να μην έχουμε προβλήματα μετά την περίοδο αυτή. Βλέπουμε τώρα ότι έχουμε ε, τέτοιου είδους επιπτώσεις. Η χώρα μου που έχει παγώσει προς αυτήν ε, η πληρωμή έχει υποστεί σημαντικότατο πλήγμα. Ναι, πράγματι είναι ένα πολύ καλό μέσο αυτό πρέπει να ομολογήσω για να αναγκαστεί μια χώρα να συμμορφωθεί με όλα τα κριτήρια και μηχανισμούς που πρέπει να ισχύουν. Όμως ταυτόχρονα στη Βουλγαρία έχουμε μια οικονομική κρίση και ενεργειακή κρίση που πλήττει τη χώρα πραγματικά οξύτατα και θα ήθελα να διασφαλίσω και να πω στην Επίτροπο ότι το ίδιο ε, αναφέρθηκε και ε, προηγούμενα ότι δηλαδή η χώρα μας έχει ήδη υιοθετήσει τα αναγκαία μέτρα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Έχουμε ένα νέο μηχανισμό για την διαχείριση και αντιμετώπιση ε, προβλημάτων ε, και διαμόρφωση των ελέγχων και αυτά τα οποία προαναφέρθηκαν μπορώ να πω ότι όλα έγιναν, όλα έγιναν όπως ε, απαιτούντο εμπρόθεσμα και νόμιμα και νομότυπα. Θέλω να δηλώσω την βούληση να ε, προσέλθουν εδώ εκπρόσωποι της κυβερνήσεως μας να εισακουστούν, να εκφράσουν τις απόψεις τους ε, ώστε να αναφερθεί ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για κράτη-μέλη σαν το δικό μας να είναι πραγματικά ισότιμοι εταίροι ισότιμοι εταίροι ώστε να μπορέσουν να υπερβούν, να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα και να συμμορφωθούν με όλα τα κριτήρια για να εφαρμοστούν όλες οι διαδικασίες, οι διεργασίες προς το συμφέρον των πολιτών μας πάντα. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ, μιλάμε βέβαια για την απαλλαγή του 2007. Το έχω πει ήδη αρκετές φορές. Εντάξει, μπορείτε να πείτε κάποια πράγματα για το 2008, αλλά έχουμε ακόμη μερικούς ομιλητές και μετά υπάρχει και ο Επίτροπος περιμένει απ' έξω. Σας παρακαλώ να το σκεφτείτε. Και υπάρχουν αρκετοί ομιλητέ που πρέπει να πάρουν το λόγο. Εντάξει, δεν θέλω να διακόψω κανένα, αλλά ε, δυστυχώ έχουμε και κάποια ευθύνη. Ο κύριο Γκαρίγκα, εν πάση περιπτώσει. Ε, Θα είμαι πανσύντομο, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα έγκριση τη διαχείριση είναι μια δυναμική διαδικασία. Οι πράξει του παρελθόντο προδικάζουν το ε, παρόν ή μπορεί να επηρεάσουν τη διαχείριση της επόμενης χρονιάς. Λοιπόν, θέλει να κρατήσει μία σκληρή στάση η επίτροπος, έτσι τουλάχιστον μας λέει, τη συγχαίρω γι' αυτό. Στα πρώτα χρόνια αυτής της ε, κοινοβουλευτικής θητείας γινόντουσαν πάρα πολλά σχόλια σχετικά με απάτες ενώ σήμερα μιλάμε απλώς για παρατυπίες ή ασυμβατότητες με την κοινοτική νομοθεσία κυρίως όσον αφορά στην ε, σύναψη των εθνικών συμβολέων. Δηλαδή πλέον έχουμε υπησέλθει στη λεπτομέρεια της διαχείρισης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι βελτιώθηκε η ποιότητα και της δαπάνης και του ελέγχου. Τώρα, ρωτώ, σχετικά με το πακέτο για της Κομισιόν για την αντιμετώπιση οικονομικής ε, ε κρίσης. Η χρήση των διαρθρωτικών ε, ταμείων χρήση των προκαταβολών και των ενδιάμεσων πληρωμών από το Ταμείο Συνοχής. Ένα από τα πιο ισχυρά μέσα που έχει η Κομισιόν για να βελτιώσει τον έλεγχο της διαχείρισης των διαφορετικών ταμείων είναι το να παρακρατά ορισμένες από τις ενδιάμεσες πληρωμές των κρατών μελών που θεωρεί ότι δεν πρέπει να δοθούν για λόγο παρατηρίας. Τώρα, στο μέλλον θα λαμβάνεται υπόψη αυτή η αντίφαση για παρακράτηση των ενδιαμέσων πληρωμών διότι υπάρχουν ακόμα κράτη-μέλη τα οποία έχουν ποσά παρακρατημένα από την Κομισιόν και δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Πολύ σύντομη απάντηση. Πρώτα απ' όλα διασφαλίζουμε αποκινούμε όλα τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή ότι τα συστήματα τα οποία βρίσκονται λειτουργία θα είναι αντικείμενο συμμόρφωση από όλου. Δεν θα υπάρξουν ενδιάμεσε πληρωμέ μέχρι ότου να συμβεί αυτό. Σημειώνουμε καλή πρόοδο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι για την περίοδο 2007-2013 τα κράτη-μέλη να αρχίσουν πραγματικά να χρησιμοποιούν τα κονδύλια τα οποία του δίνονται ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή προκαταβολών. Δεν βλέπω λοιπόν πραγματικά να υπάρχει κάποια αντίφαση οπωσδήποτε είναι προς και προς το συμφέρον επίσης των κρατών μελών ώστε στο τέλος τέλος να μην υπάρχουν άλλες διαδικασίες ελέγχων με ε, απαιτήσει ανάκτησης κτλ. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Γκρέσλα, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε που μου δίνετε την δυνατότητα να παρέμβω. Στην αρχή και όλα στις παρέμβασή μου είχα μια κακή αρνητική συνείδηση διότι δεν είμαι εγώ ελέγκτρια και προσπαθούμε από κοινού μια πολιτική για την πολιτική ολοκλήρωση στην Ευρώπη, στις περιφέρειες να λειτουργήσει σωστά και να επιτευχθεί. Όμως είμαι ωστόσο πάλι εκείνοι που από τους φορείς των προγραμμάτων, από τις ε, κοινότητες, τους δήμους, τις περιφέρειες, οι πρώτοι είμαι που παίρνω τα μηνύματα γιατί τα δυσχεραίνουμε όλα για εκείνους ώστε να μην αξίζει πια τον κόπο να ξεκινούν τέτοια προγράμματα για την υλοποίηση αυτών των στόχων και εκεί έχουμε και πολύ έντονη τη συνιστόσα των ελέγχων. Γι' αυτό είμαι ευγνώμων στον κύριο Οντή ότι το θέμα της απλούστευσης το έθιξε και το κάλυψε με αυτόν τον τρόπο την τελευταία εβδομάδα και του τελευταίους μήνες ασχολούμαι πάρα πολύ σε βάθος έντονα με αυτή την αντίφαση. Θέλουμε στις περιφέρειες να ακολουθηθεί μια πολιτική με τέτοιο τρόπο ώστε τα χρήματα των φορολογουμένων, τα κονδύλια που παρέχουμε να παρέχονται με τον καλύτερο τρόπο. Είναι αντίφαση αυτό το εγχείρημα επειδή στις ιδέες μας που μας εμπνέουν το δυνατόν όλα να τα καθορίσουμε επακριβώς πώς κάθε δεκάρα θα μπορεί να θα επιτρέπεται να δαπανάτε έχουμε φτάσει τόσο μακριά και έχουν πάει τόσο μακριά ώστε είναι πάρα πολύ δύσκολοι οι κανόνες, περίπλοκοι. Χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο χοντρό εγχειρίδιο για να μπορεί κανεί να τα κατανοήσει, να επεξηγηθούν και δεν απλουστεύονται αυτά από τη γραφειοκρατία που επιπλέον σε εθνικό επίπεδο και περιφερειακά και τοπικά επιβαρύνουν όλα αυτά. Γι' αυτό κατεπίγουσα παράκληση να έχουμε πιο απλούς, πιο διαφανεί κανόνε που θα μπορούν να γίνονται κατανοητοί άμεσα και όχι παρερμηνεύοντας κανόνε να καταλήγουμε σε σφάλματα. Από την άλλη τώρα πλευρά θα ήθελα για άλλη μια φορά να καταστήσω απόλυτα σαφές 11% ποσοστό σφάλματος είναι υπερβολικό. Θα ήθελα οπωσδήποτε να μειωθεί αυτό. Από την άλλη πλευρά 11% σφάλμα δεν σημαίνει 11% απάτες, περίπτωση απατών. Αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο εισηγητής με κάθε σαφήνεια κάθετα το ανέφεραν. Δηλαδή αντιστρέφοντας τους όρους πάλι σημαίνει δεν είναι κάθε ένας που κάνει λάθος ένας απατεώνας. Απευθύνω έκκληση λοιπόν σε εσά αγάπη αγαπητοί αξιότιμοι συνάδελφοι να μην είμαστε ισοπεδωτικοί ε, με, αυτό, με μια τέτοια προσέγγιση και στις περιφέρειες ή και στην Ευρωβουλή να μην με το ψαλίδι κόβουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να λέμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμήσουμε τους απαταιώνες. Όπου γίνεται δουλειά γίνονται σφάλματα, γίνονται λάθη και ακριβώς σε έναν τομέα όπου η Ευρωβουλή θέλει να προαγάγει ιδιαίτερα την καινοτομία για παράδειγμα για να έχουμε αηφόρες επιπτώσεις στη διαθροτική πολιτική, στην καινοτομία και καινοτόμα δράση για παράδειγμα να το δούμε και αυτό εμπεριέχεται έτσι και υπάρχει και υψηλότερο ποσοστό σφάλματος εκεί. Είναι λογικό και συνεπές αυτό. Πρέπει πρώτα να δοκιμάσουμε κάτι, να δούμε αν δουλεύει, αν λειτουργεί καλά. Αν υψηλότερα ποσοστά σφάλματος οδηγούν ώστε ένα συνολικό πρόγραμμα να παγώνει και να μην πληρώνουμε πια προκαταβολές επειδή αυτό προβλέπεται από τους κανόνες και δεν επιτρέπεται να υπερβούμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό σφάλματος, ε, πού θα φτάσουμε πια ένα κράτος μέλος ή μια περιφέρεια θα ακολουθεί μόνο με τις ε, παλαιές μεθόδους που γνωρίζουν ένα πρόγραμμα ή ένα σχέδιο για την, ένα διοικητικό κέντρο ή για τη δημιουργία ενός δρόμου, μιας οδού ή θα εξηγιένεται κάτι με μια βιομηχανία. Θα γίνονται πράγματα όμως τα οποία δεν μας πάνε πολύ πιο πέρα, πολύ πιο μακριά πρέπει μεταξύ εκείνων που διαθέτουν τα κονδύλια και εκείνων που θέλουν να εφαρμοστεί μια πολιτική και εκείνων που πρέπει και μπορούν να κάνουν τους ελέγχους να βρεθεί ένα, μια κοινή βάση και ελπίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα παραμείνει εκεί στάσιμη αλλά θα συνεχίσει παραπέρα και στο θέμα της απλούστευσης. Συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Ντούχον, έχετε τον λόγο παρακαλώ. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Με το υψηλό ποσοστό σφάλματο που έχουμε απέναντί μα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά επίση και με ανεπάρκεια για την ε, βεβαιότητα όσον αφορά αυτά τα σφάλματα. Πού έγκυται το πρόβλημα. Οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ, ιδιαίτερα η πολιτική συνοχή και η πολιτική γεωργία ε, που ακολουθούν οδηγούν στην καταβολή πληρωμών σε ύψο ε, εκατομμυρίων ετήσια πολύ ψηλά αυτά τα ποσά. Μπορώ να τολμήσω και να πω ότι είναι ανεξέλεγκτα και ανέλεγκτα υπό την προϋπόθεση πάντα ότι δεν ε, θα είναι ε, διαρκώς, δεν θα διευρύνονται διαρκώς ε, οι έλεγχοι όσον αφορά το ελεγκτικό συνέδριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό το σφάλμα. Απευθύνει έκκληση για την μείωση του ποσοστού σφάλματος. Ζητά να υπάρξει απλούστευση των συστημάτων ε, της προσέγγισης. Δεν πρέπει να παραμείνουμε στάσιμοι. Το λογικό συμπέρασμα βλέπω να είναι ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε επιθεμάτων αρχής στην ευρωπαϊκή πολιτική να την μειώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε θα μειώνονται οι πληρωμές ετήσια. Θα με ενδιέφερε να ακούσω ποια είναι η άποψη της Επιτρόπου για αυτήν την πρόταση. Ευχαριστώ. Ναι, θα μας απαντήσετε. Οπωσδήποτε θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τον αριθμό των πληρωμών ανά έτος, αλλά έχουμε ένα σύστημα ομαδοποίησης το οποίο θα πρέπει να μας βοηθήσει. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω σαφώς, ίσως στο μέλλον να μπορεί να βοηθήσει δήμους και λοιπούς. Εάν μπορούν να κάνουν ε, ομαδικά τις αιτήσει τους ε, για μικρά έργα προς την Κομισιόν. Αυτό είναι και στις παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Έτσι ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία η διοικητική χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μειώνεται ο έλεγχος των ε, δαπανών. Μάλιστα, για τους συναδέλφους που δεν είχαν χτες το χρόνο να πάσουν χτες, νομίζω ότι χρησιμοποιήσαμε ένα αρκετά μεγάλο τμήμα του χρόνου για να συζητήσουμε το ανεκτό ε, σφάλμα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εμείς δεν είμαστε κατά του να δίδονται τα χρήματα, απλά να δίνονται λογικά. Κύριε Φασάκα, έχετε τον λόγο. Ναι, θα... είμαι σύντομος καθώς οι προλαλήσαντες το ανέφεραν ε, το θέμα το οποίο ήθελα να θίξω. Παρόλα αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για το ότι ε, απαντάει όλες τις ε, ερωτήσεις μας εδώ πέρα και είναι στην διάθεσή μας. Είναι καλό να βλέπουμε πώς θα οδηγηθούμε σε καλύτερη συνεργασία. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, έχετε δίκιο πως ε, τελικά προεδρε εχετε δει και όπω τελικα μιλαμε για την απαλλαγή του 2007, αλλά στόχος μας εδώ πέρα δεν είναι πάντα να κρίνουμε μόνο το παρελθόν, αλλά να μέσω αυτού να εξετάζουμε τις μεθόδους και να βελτιώνουμε τη συνεργασία για το μέλλον. Γι' αυτό η ερώτησή μου, η τοποθέτησή μου αν θέλετε, και είναι κάτι το οποίο αναφέρθηκε ήδη και απαντήθηκε από τους συναδέλφους πώς βλέπετε την σημερινή κατάσταση που είναι μια κατάσταση ανάγκης στην Ευρώπη πολλά στις περισσότερες χώρες πλέον είναι σε δινή θέση πώς βλέπετε θα γίνει αυτός ο τετραγωνισμός του κύκλου δηλαδή να γίνουν αυτές οι πληρωμές πιο εύκολα με λιγότερη γραφειοκρατία γρηγορότερα χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα αυξηθεί ο κίνδυνος ε, σφαλμάτων και χωρίς να διακινδυνεύσει η εξοπιστία αυτών των πληρωμών και κατόπιν ένα ακόμα ερώτημα αν θέλετε το απαντάτε τώρα αν όχι κάποια στιγμή στο μέλλον ποια συγκεκριμένα βήματα σκοπεύετε να κάνετε και στο μέλλον βεβαίω, ε, όπως ε, είπε και η κυρία Κούψεβα για να έχουμε πραγματικά συγκεκριμένη πρόοδο πρώτον για τη μείωση της γραφειοκρατίας γρηγορότερες πληρωμές β, νέα θέματα, νέοι στόχοι που θα πρέπει να συμπεριληφθούν που δεν υπάρχουν ε, αυτή τη στιγμή και δεν προωθούνται από την Ευρώπη και ένα τελευταίο ερώτημα, κάτι που διάβασα στον τύπο είναι γεγονός πως για τη Ρουμανία οι προκαταβολές ε, αυξήθηκαν από το 3 στο 4% ε, τι γίνεται έγινε αυτό μετά από μια συμφωνία με το Κοινοβούλιο και εάν ναι αυτό ισχύει γενικά ή διαφέρει από χώρα σε χώρα βεβαίως αυτό δεν σχετίζεται με την απαλλαγή αφορά το μέλλον Πολύ σύντομα, επειδή είναι τεράστιο θέμα αυτό και για την κρίση, για την χρήση αυτών των πολιτικών ως την μεγάλη επένδυση, κίνητρο επενδύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτικών και έτσι αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως την ελαστικότητα που υπάρχει στη διάθεσή μας και αποφασίσαμε να επεκτείνουμε την επιλεξιμότητα για τη χρηματοδότηση 2000-2006 και για, όπως και φέτος να απλουστεύσουμε σε μεγάλο βαθμό όλα τα μέτρα πολιτικής που συνεισφέρουν υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη ε, ρευστών, την έλλειψη χρημάτων σε αυτόν τον τομέα ώστε να υπάρχει δυνατότητα και πρόσβαση σε, σε πιστώσεις ε, για αυτές τις επιχειρήσεις και να υπάρξει μεγαλύτερη χρηματοδότηση και στην αγορά στην αρχή αυτής της διαδικασίας κιόλας και όχι στο τέλος της διαδικασίας πρόημα δηλαδή. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τις επιπρόσθετες προκαταβολές ε, προεξοφλητικά και τις πληρωμές που υιοθετούν τα κράτη-μέλη και τώρα υπάρχει η ανάγκη να δώσει σύμφωνη γνώμη, να εγκρίνει η Ευρωβουλή. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τα 15 παλαιότερα κράτη-μέλη που παίρνουν επιπλέον 5% και τα 12 προηγού παλαιότερα κράτη-μέλη που, παίρνουν, που παίρνουν επιπλέον 2% και για την βοήθεια υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνικών και την υποστήριξή τους. Επίσης αποφασίσαμε ότι και μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αυτή η πολιτική έχει ήδη δώσει αποτελέσματα και έχει δώσει αντιδράσεις ε, σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές για παράδειγμα και τι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρησιμοποιούμε αυτή τη δυνατότητα για να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις σε σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, τις κλιματικές αλλαγές, ε, την δημιουργία ανάκαμψης. Με αυτές τις πολιτικές δρούμε υπάρχουν ευκαιρίες μέσα στο πλαίσιο τη της νέας βιομηχανικής επανάστασης εδώ. Η απλούστευση, η εξαπλούστευση και η επιτάχυνση εξεράχυνση της ε, διάθεσης των κονδυλίων που θα είναι διαθέσιμα με κάθε σεβασμό φυσικά προς το σύστημα δημοσιονομικών ελέγχων ευελπιστούμε ότι θα μπορέσει να βοηθήσει την ευρωπαϊκή, να βοηθήσουν την ευρωπαϊκή οικονομία όλα αυτά τα μέτρα να εξέλθει από αυτή την κρίση. Τέτοιου είδους επενδύσεις είναι αυτές που χρειαζόμαστε σήμερα για να αναζωογονήσουμε την ε, δυναμική της οικονομικής ζωής και πρέπει να έρθει από κάτω από το τοπικό επίπεδο ακολουθώντας αυτές τις πολιτικές είναι λοιπόν χρήσιμες αυτή στιγμή και ελπίζω ότι η απλούστευση, η εξαπλούστευση θα διευκολύνει και τα πράγματα. Ευχαριστώ. Okay, Ωραία, ευχαριστούμε. Προσέξτε, σας παρακαλώ να μην βρίσκεται κανείς εδώ πέρα σε αυτή τη θέση σε δύο χρόνια και να λέει Θεέ μου ποιος να το ήξερε και να έχουμε τέτοιες, τέτοιες ε, εκπλήξεις όχι μόνο στις Βρυξέλλες αλλά και αλλού και να με συγχωρείτε που το λέω. Λοιπόν, Κυρία Λοκούρτου, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα. Ε, ε, Θα ήθελα να εκφράσω την θετική μου εντύπωση για την παρουσίαση της Επιτρόπου Υμπνεχ και στα πρώτα αποτελέσματα της εφαρμογής του σχεδίου δράσης. Είναι πολύ θετικό το πώς εφαρμόζεται και επίσης σέβεται και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι της Επιτροπής μας και του Κοινοβουλίου η υλοποίηση του σχεδίου δράσης είναι θεμελιώδες, θεμελιώδης για να περιορίσουμε και το περιθώριο λάθους στα διαρθρωτικά ταμεία. Και το θέμα της ε, ανάκλησης ε, πληρωμών ε, και οι διορθώσεις που μας ανέφερε η Επίτροπος μας δείχνει ότι έχουμε μπει σε καλό δρόμο. Μίλησαν πολλοί συνάδελφοι γι' αυτό αλλά και η ίδια η Επίτροπος για την ανάγκη της απλούστευσης των διαδικασιών και των κανόνων. Αυτό είναι θεμελιώδες για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα λάθη και να δαπανούμε καλύτερα τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων. Και το ελεγκτικό συνέδριο διαπίστωσε αυτή τη βελτίωση. Τώρα, μόνο έξι προγράμματα στα 16 θεωρούνται αναποτελεσματικά Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα που κάναμε προς τα μπρος. Ελπίζω ότι θα έχουμε μία πιο αποτελεσματική σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και Κομισιόν. Όσο πιο ισχυρά οικοδομούμε εμείς αυτή την σχέση αλληλεπίδρασης, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι και το μέσο το οποίο δίνουμε εμείς στα κράτη-μέλη. Λοιπόν, ρωτώ την Επίτροπο, τι προβλέπει για το 2009 το σχέδιο δράσης. Και τελευταίος ο συνάδελφος Ούλμπριχτ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Okay, thank you. First, uh, uh, two remarks and two questions. Ε, δύο σχόλια, μία ερώτηση. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι μιλάμε για το 2007. Μιλάμε... Είμαστε στην Επιτροπή Ελέγχου του Υπερπολογισμού. Πρέπει να το πούμε αυτό. Συγκεκριμένα και για τις άλλες επιτροπές, γιατί μιλάμε συγκεκριμένα για τα συμπεράσματα του 2007 δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, για, να μιλάμε για το 2008, είναι τελείως διαφορετικά τα, τα πράγματα. Ποια, να λέμε ποια ήταν η τάση του 2007 χωρίς το σχέδιο δράσης, γιατί το σχέδιο δράσης ήταν μετά το 2007. Οπότε το θέμα ήταν ποια ήταν η τάση το 6 και το 7, γιατί το σχέδιο δράσης είναι μια απάντηση σε αυτό. Δεύτερη παρατήρηση. Στην ε, Επιτροπή μας ε, συζητάμε ακόμα τι, τι γίνεται σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και τα λάθη, τα ασφάλματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη σχέση ανάμεσα στα ασφάλματα και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μετά από αρκετά χρόνια, γιατί δεν θέλω να πω πως τα περισσότερα ασφάλματα είναι καλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά είναι γεγονός πως ε, η χειρότερη πολιτική είναι το αποτέλεσμα των σφαλμάτων. Μπορούμε να έχουμε και πολλά σφάλματα και καλή πολιτική ταυτόχρονα. Αυτό είναι πολύ βλοκό το ζήτημα γιατί υπάρχουν διαφορετικές προοπτικές. Αν μιλάμε για ένα έτος ή για πολλά και βέβαια όλα αυτά τα εξετάζουμε κάποια χρόνια αφού έχει λήξει η πολιτική. Τι γίνεται με την πολιτική όμως, γιατί ακούμε τα συμπεράσματα εντός του Κοινοβουλίου πως λόγω των διαδικασιών, λόγω των σφαλμάτων, ας την ξεχάσουμε αυτή την πολιτική. Ε, ε, ε, να με συγχωρείτε, αλλά αυτά είναι τρελά πράγματα. Μιλάμε για τι διαδικασίε, μιλάμε για τα σφάλματα, αλλά το, το πρόβλημα τη αποτελεσματικότητα τη πολιτική είναι τελείω διαφορετικό. Τώρα, δύο ερωτήσει. Πρώτον, υπάρχει ορατός κίνδυνος σε επίπεδο δικαιούχων. Αυτή η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να οδηγήσει σε περισσότερο έλεγχο και όχι σε λιγότερο. Όχι απλοποίηση, αλλά περισσότερο έλεγχο. Το ερώτημα είναι τι θέλει να κάνει η Κομισιόν για να μην οδηγηθούμε σε περισσότερο έλεγχο στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά σε καλύτερο έλεγχο, γιατί το πρόβλημα το βλέπουμε εδώ πέρα στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βλέπουμε τους τύπους των ελέγχων. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Λένε πω ένα τύπο ελέγχου γίνεται τρει φορές. Οπότε να μην έχουμε τέσσερι ελέγχου, αλλά 11, 12, γιατί όλοι φοβούνται. Οπότε το ζήτημα δεν είναι όχι περισσότερου ελέγχου, αλλά καλύτερου. Και το άλλο ερώτημα του κύριου Ντεμπλάζια γιατί στη συζήτησή μας βλέπουμε πως υπάρχουν διαφορετικά πύχη κριτήρια επιλεξιμότητας ε, στα κράτη-μέλη και διαφορετικά στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι το οποίο είναι επιλέξιμο εντός της χώρας δεν είναι επιλέξιμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ερώτημα είναι τι ε, θεωρεί η Κομισιόν ότι είναι το ποσοστό αυτού του προβλήματος ε, ως ε, ποσοστό των λαχών. Δηλαδή να μην υπάρχει πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο, αλλά να είναι το ίδιο πράγμα μη επιλέξιμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε χάνονται οι δικαιούχοι και παγιδεύονται. Δεν έχω απάντηση βεβαίω για το τι πρέπει να γίνει. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τέλο πάντων δεν είναι εύκολο αυτό. Τελευταία παρατήρηση. Το ping-pong είναι ενδιαφέρουσα διαδικασία. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και στην Επιτροπή μα. Ακόμα και αν δεν είναι πάντα η γρηγορότερη. Ναι. Πρέπει, πρέπει επίσης να, μάθουμε να είμαστε και λίγο πιο σύντομοι. Ελπίζω αυτές οι δύο ερωτήσεις να μπορέσουν να απαντηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακριβώς μια και εδώ κάνουμε λόγο για το θέμα του αποδεκτού κινδύνου tolerable risk, συνάδελφε Ολμπρίστ. Πήρα κάποια στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επειδή γίνεται λόγος για ελέγχους και τέτοια συχνότητα, τα στοιχεία που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι λένε, Περιφερειακό Ταμείο 0,7%, 0,7%, Κοινωνικό Ταμείο 0,8%. Δηλαδή εκπληκτικά χαμηλά αυτά τα αριθμητικά μεγέθη. Θα έπρεπε ή θα μπορούσαν να είναι πολύ ψηλότερα. Εντάξει, αυτό είναι το έτοιμά μας, αλλά να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Αυτά πληροφοριακά. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτέ τι δύο ερωτήσει του συναδέλφου Όλμπριχτ υπάρχουν κάποιε παρατηρήσει για να, να απαντηθεί. Σύντομα παρακαλώ. Σύντομα. Γνωρίζοντα ε, ότι για αυτές τις ερωτήσεις που τίθενται και για την απάντησή τους στεναρά πιστεύουμε ότι με αυτή τη συζήτηση φυσικά φυσικά υπάρχουν πολλές επιπτώσεις ή συμπεράσματα που μπορούν να συναρθούν και εκτός αυτής τη αιθούση και εκτός Βρυξελών. Όμως η πρόθεσή μας, η δική μας κατανόηση του νοήματος αυτής τη συζήτηση είναι ότι όλοι θέλουμε να υπάρξει ένα καλύτερο σύστημα που θα δημιουργηθεί, καλύτερο όσον αφορά τη διαχείριση, καλύτερο όσον αφορά την λογοδοσία, καλύτερο όσον αφορά επίση και τα αποτελέσματα τα οποία θα δίνει με συγκεκριμένους όρους χειροπιαστά. Ελπίζουμε ότι αυτή η συζήτηση θα βοηθήσει να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχων και ελεγκτικό Αποκινούμε τις εθνικές ε, ε, πιστοποίησεις και δηλώσεις. Κινούμαστε προς μια κατεύθυνση ε, αλλά δεν βλέπουμε, δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα και σε σχέση με κάποια κράτη-μέλη έχουμε συγκεκριμένες καταστάσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση ε, και των ε, ε, παρατυπιών και όσον αφορά τις αλλαγές που είναι πάρα πολλές και σε σχέση και με τις εθνικές πιστοποίησεις ή δηλώσεις. Έχουμε φτάσει σε μια κριτική μάζα που θα μπορέσει να βοηθήσει στο τέλος να μειωθεί το κόστος των ελέγχων και οι έλεγχοι θα γίνουν και πιο υπεύθυνοι θα έλεγα και πιο αποτελεσματικοί. Διότι θεωρώ πραγματικά ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι η επίπτωση που θα έχει αυτή η πολιτική στις αλλαγές ε, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίας. Πράγμα που καμιά φορά το ξεχνάμε όταν συζητάμε. Διότι συζητούμε τις περισσότερες φορές αυτές τις πτυχές αλλά δεν συζητάμε την άλλη όψη αυτού του νομίσματος αυτής της πολιτικής και τις άλλες ε, παραμέτρους. Τώρα για τη δεύτερη ερώτηση δεν γνωρίζω την απάντηση, δεν μπορώ να την ε, ε, αναφέρω σε αριθμητικό μέγεθος. Όμως σε σχέση με το σύστημα δεν έχουμε τόσους ελέγχους σε σχέση με τις εθνικές δημόσιες πολιτικές τέτοιου είδους, τέ, τέτοιου είδους ελέγχους δηλαδή. Υπάρχει αυτή η πτυχή της πολιτικής που πρέπει και αυτή να ληφθεί υπόψη και να συμπεριληφθεί τον τρόπο δηλαδή που πρέπει να πορευτούμε προς το μέλλον που θα ήταν να ληφθεί και αυτό υπόψη, να ενταχθεί και αυτό και σε ένα σύστημα το οποίο θα υιοθετηθεί να μπορεί να καλύπτεται αυτή η πτυχή υπό τις εθνικές πολιτικές συνδυάζοντας την ευρωπαϊκή διάσταση και την εθνική διάσταση σε μία αναπτυξιακή πολιτική ενιαία. Αυτά είναι όμως θέματα που εκκρεμούν ακόμα ή μένουν ακόμα ανοιχτά. Μπορεί το ελεγκτικό συνέδριο να προσπαθήσει να απαντήσει με κάποιες παρατηρήσεις ακριβώς για την τελευταία αυτή παρέμβαση του κ. Όλμπρεκτ. Παρακαλώ κυρία. Ευχαριστώ. Ήθελα να σχολιάσω μία πτυχή το ερώτημα που κάνετε. Δηλαδή αν είναι περισσότερα τα λάθη σημαίνει ότι είναι χειρότερη η πολιτική. Εάν δείτε Αν δείτε το τι γίνεται σε σχέση με τις διορθώσεις στα ανατολικά κρατημέλη και ότι υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός για να προσελκυστούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και αν υποθέσουμε πως υπήρχε ένα έργο το οποίο είχε έρθει πρώτο αλλά ήταν ε, λανθασμένο και αντικαταστάθηκε από ένα άλλο γιατί ε, έπρεπε και γιατί ο χρόνος πίεζε κτλ. Ναι, οπωσδήποτε έχει και αρνητικό αποτέλεσμα στην πολιτική. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την μακροσχελή αυτή και αναλυτική συζήτηση. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή, την ε, Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τελειώνουμε με αυτό το μισό σημείο. Κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα για να αλλάξουμε θέσεις και θα συνεχίσουμε με τον Επίτροπο, τον κύριο Ποτότσνικ.